Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε φορτωμένη ημερήσια διάταξη σήμερα. Προτείνω να αρχίσουμε, οι άλλοι συνάδελφοι θα έρθουν αργότερα. Εμείς έχουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 26ης Μαΐου, 14ης, 15ης Ιουνίου, 30 Ιουνίου, 12 Ιουλίου που είναι στη διάθεσή σας και αν δεν έχετε καμία αντίρρηση θα τα εγκρίνουμε. Λοιπόν, έχουμε τρεις περιόδους ε, σήμερα στη συνεδρίασή μας. Θα έχουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων στην έκθεση του συναδέλφου και αντιπροέδρου Κρίστοφ Λίζεκ για τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα. Μετά θα έρθει ο Αλέν Λερουά, ο οποίος ε, ε, έχει πλέον ε, ολοκληρώσει τη θητεία του στον ΟΕ στη διεύθυνση του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων και μετά θα έχουμε τον κύριο Κασάλμι. Σάλμη, για τον ρόλο και τα καθήκοντα του κέντρου επιχειρήσεων. Επίσης, έχουμε ένα σημείο επικαιρότητα το οποίο είχαμε στην ημερήσια διάταξη όπως το θύμισε και ο κύριος Ποπόβς και χτέ το συζήτησαν οι Υπουργοί Άμυνας. Θα το ξανασυζητήσουν στην επίσημη συνεδρίαση στις 30 Νοεμβρίου οι Υπουργοί Άμυνας και με αυτό το θέμα έχουμε κάτι το οποίο βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο των ανησυχιών των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, ε, ο, οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Άμυνα εργάζεται επίσης ε, στον ε, τομέα του pooling and sharing και ο Λίσεκ εργάζεται για τη διατύπωση των προτάσεων. Κριστόφ, Χωρίς να περιμένω παραπάνω σου δίνω το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ανησυχώ Α, να, υπάρχει διερμηνία. Βεβαίως και υπάρχει διερμηνία. Ανησυχώ λοιπόν έλεγα διότι έχουμε την Κυριακή εκλογές στην Πολωνία και πρέπει να ασχοληθώ με θέματα εντελώς διαφορετικά. Φυσικά, έχουμε και όλη τη δραστηριότητα της Πολωνικής Προεδρίας και όπως είπε και ο κύριος Ποπόφσκι, η Πολωνική Προεδρία θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας να τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών δομών. Στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας εδώ και καιρό συζητάμε για τις προτάσεις της Πολωνικής Προεδρίας σχετικά με την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Όπως είπε και ο πρόεδρος, η υπάρχει μία τεράστια σύμπτωση απόψεων μεταξύ αυτών που λέμε εμείς και αυτών που λένε οι εμπειρογνωμονές που γνωρίζουν πολύ καλά τις δομές του ΟΙΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ δεν θα σας διαβάσω εδώ όλη την έκθεση, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τη γνωρίζετε πολύ καλά την έκθεση την έχετε μπροστά σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της υποεπιτροπής που είχαν την ευγένεια να μου υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους. Μόλις καταστεί δυνατόν θα σας στείλω ένα σχέδιο έκθεσης και αυτό το το οποίο σας έχω υποβάλει σήμερα λαμβάνει υπόψη σημαντικές παρατηρήσεις των μελών της Υποεπιτροπής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ανοιχτό προς συζήτηση, προς συνδυασμό, προς όλα. Δεν πιστεύω ότι είμαι παΐων στο θέμα. Αυτή η έκθεση είναι πάντοτε ανοιχτή σε οποιαδήποτε τροποποίηση για να μπορέσει να συμπεριλάβει την κοινή γνώμη της Επιτροπής μας. Αρχίζοντας να σας πω ότι με τους συμβούλους μου και με την γραμματεία είχαμε συναντήσεις με τους εμπειρογνώμονες, βασιστήκαμε και στην ακρόαση και αυτά τα και αυτά, όλα αυτά αποτελούν την τεκμηρίωση των όσων θα σας προτείνω. Τις τελευταίες εβδομάδες είχαμε ε, συναντήσεις με όλους όσους ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ασχολούνται με θέματα άμυνας και ασφάλειας. Συζητήσαμε με, με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας, Ώρες και ώρες συζητήσαμε. με εμπειρογνώμονες και ειδικού, διαβουλευθήκαμε και την Πολωνική Προεδρία. Και όλα όσα μας είπανε τα έχω συμπεριλάβει στην έκθεση μου και ελπίζω ότι θα τα συμμεριστείτε κι εσείς. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό πριν ξεκινήσουμε με την ανάλυση των σημείων κλειδί αυτής της έκθεσης ότι η κατάσταση σήμερα στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη είναι παρόμοια συζητώντας με την εκπρόσωπο, την είπατε εκπρόσωπο εξωτερικών της Ένωσης αλλά και με τους εκπροσώπους των κρατών μελών όλοι είπανε ότι χρειαζόμαστε αναδιαρθρωτικά μέτρα γρήγορα και αποτελεσματικά. χρειαζόμαστε κοινέ δράσεις. Και τώρα έρχομαι εδώ πια στο περιεχόμενο της έκθεσής μου. Και λέω ότι σήμερα επίγουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, διότι η οικονομική κρίση φύγει σχεδόν όλα τα μέλη των κρατών μελών. Ε, συγγνώμη, όλα τα κράτη-μέλη. και πολλά κράτη-μέλη λόγω αυτής της κρίσης προχωρούν σε περικοπές στον προϋπολογισμό άμυνας. Αλλά άμα δείτε τι γίνεται γύρω μας και τους τελευταίους μήνες, ε, Λιβύη, Ιράν κλπ, αυτές οι περικοπές ε, παίρνουν μια άλλη διάσταση στο τωρινό πλαίσιο. Συζητήσαμε με τους ε, Βρετανούς ε, εμπειρογνώμονες. Η Μεγάλη Βρετανία σε σύγκριση με την Πολωνία έχει στη διάθεσή της έναν εντυπωσιακό προϋπολογισμό για θέματα άμυνας. Και λένε ότι για να συνεχίσουν τη δράση τους οι Βρετανικές δυνάμεις ε, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ πρέπει να εξαντλήσουν τα κονδύλια τα οποία έχουν στη διάθεσή τους. Αυτά δηλαδή τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους δεν αρκούν για τη συνέχιση της δράσης τους. Αναφέρω εδώ το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας η οποία έχει πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό άμυνας έναντι της Πολωνίας. Στην έκθεσή μου τονίζω και κάτι άλλο. Αν θελήσουμε να υπολογίσουμε το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού άμυνας των κρατών μελών, θα καταλήγαμε σε ένα πολύ σημαντικό ποσό, 200 δις ευρώ. Αν τον συγκρίνουμε όμως αυτόν τον προϋπολογισμό με τον προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, οχριούμε διότι ο προϋπολογισμός μας είναι τρεις φορές μικρότερος από τον αμερικανικό προϋπολογισμό. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Διότι τις μεγαλύτερες δαπάνες τις υποστηρίζουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αυτό είναι και το σημείο, το σταυρικό σημείο της έκθεσης που σας υποβάλλω. Οι εμπειρογνώμονες της έντα λένε ότι αυτά τα 200 δις είναι παραπάνω από ότι αυτά που ξοδεύουν η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ρωσία, λέει ο μιλητής. οι δαπάνες για τους εξοπλισμούς αυξάνονται διότι η τεχνολογία προχωράει, οι εξοπλισμοί είναι συνεχώς πιο εξεζητημένοι. Πρέπει κατά συνέπεια να έχουμε μία κοινή συνεργασία, να έχουμε έναν κοινό σχεδιασμό να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε από κοινού για να δαπανίσουμε σωστότερα τα χρήματά μας. Διότι αυτός ο προϋπολογισμός με στενή συνεργασία θα ξοδευτεί με καλύτερο τρόπο και πιο στοχευμένα. Έχω κατά νου εδώ το pooling and sharing, αυτό που ο κύριος Ποπόφσκι χθε υπογράμμισε πολλές φορές. Το pooling and sharing είναι μία ιδέα, ένα όνειρο που έχει αρχίσει να παίρνει όμως συγκεκριμένη μορφή στις σκανδιναβικές χώρες. Και σήμερα καθίσταται κάτι παραπάνω από όνειρο, είναι πλέον ανάγκη και πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα σε μεγάλη κλίμακα, όχι σε μικρέ, μόνο σε μια μικρή ομάδα χωρών. Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη φόρμουλα. Εμείς έχουμε ένα σωρό ωραία παραδείγματα πάνω στο οποία μπορούμε να βασιστούμε. Αλλά η εμβάθυνση τη συνεργασίας πρέπει να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο κύριος Ποπόφσκι εχθές ανέφερε σχέδια προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό νέο που θα συζητηθεί στην συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στο Βρόκλαβ. Ο κύριος Ποπόφσκι είπε ότι θα μπορούσαμε ε, ε, να εντάξουμε σε αυτή τη λογική τις ε, ιατρικές θεραπείες, την κατάρτιση των πιλότων, κοινή κατάρτιση. Οργάνωση, δηλαδή της διάρθρωσης των δαπανών. να αξιοποιήσουμε την δαπάνη στο maximum σε όλα τα επίπεδα. Και αν πετύχουν όλα αυτά, τότε θα ενισχυθεί και όλο αυτό το pooling and sharing. μόνο το 1% των συνολικών δαπανών για την άμυνα το αφιερώνουμε στην έρευνα και στην τεχνολογία στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για έναν επαρκέστατο ποσοστό και πρέπει να το πούμε καθαρά αυτό. Και αν η Ευρώπη θέλει να παίξει σημαντικό ρόλο ως παγκόσμιος πρωταγωνιστής, θα πρέπει να καταστήσει προτεραιότητα την τεχνολογική ανάπτυξη. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτόν τον τομέα και πιστεύω ότι πρόκειται, ε, ότι πρόκειται για έναν οργανισμό ο οποίος υποτιμάται από πολλά κράτη-μέλη. Φυσικά, σε αυτήν την έκθεση υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα ήθελα να σας αναλύσω. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε βέβαια και είμαι πια πολύ περίεργος να ακούσω τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας σε λίγο. Δεσμεύομαι να συνεχίσω τη δουλειά μου σε αυτήν την έκθεση. Τελειώνω λοιπόν με αυτές τις παρατηρήσεις και άμα έχουμε χρόνο μετά θα ξαναπάρω το λόγο στο τέλος της συζήτησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένη αυτή η έκθεση διότι εξετάζει όλες τις ε, πτυχές ε, ε, του θέματος. μέγα μέρο αφορά στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση. Αυτό το διαπιστώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ο πρόεδρος Μπαρόσο στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε αυτόν τον κοινό άξονα ως προτεραιότητα, χωρίς βέβαια να μας πει αναλυτικά τι θα πρέπει να γίνει. Αλλά εμείς θα πρέπει να καλέσουμε την Κομισιόν να μας διευκρινίσει καλύτερα τη σκέψη της για αυτήν την για τη στρατηγική, για την πολιτική όθηση που προτίθεται να δώσει. Ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κλίζεκ. Πολύ καλό το σχέδιο της έκθεσης του. Ε, συμφωνήσαμε και δικαίω ότι εδώ στην Επιτροπή θέλαμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και για τους επίκαιρους λόγους που το προκαλούν ίσως για τον τομέα αυτό η κρίση, η οικονομική κρίση να αποτελεί μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία έτσι ώστε η εμπεριστατωμένη ανάπτυξη και η συνεργασία να εδρεωθούν όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Χαίρομαι πολύ που από τους υπουργούς ακούσαμε ότι είναι και αυτοί διατεθειμένοι να το πράξουν. Βεβαίως τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι στην πράξη και συμφωνώ και με τον συνάδελφο ότι σίγουρα η υπηρεσία άμυνας θα πρέπει να αποτελέσει μια κεντρική υπηρεσία από την οποία θα συντονίζονται όλα αυτά τα θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού κτλ. Έτσι ώστε να είναι όλα τα σχέδια συμβατά μεταξύ τους και να μας οδηγούν στο να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες συνεργασίας για κοινά προγράμματα. Όπου κάνουμε ε, κάτι καλό, ε, θα μπορούσαμε ίσως να το χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Ό,τι δηλαδή έχει υπάρξει από το παρελθόν, να το βάλουμε και αυτό στο pooling and sharing. Και στον τομέα αυτό υπάρχουν ε, περίπου 330 εγκεκριμένα προγράμματα. Οπότε τώρα θα πρέπει να δούμε αν όντως όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν. Και εμείς εδώ στην ε, Επιτροπή μας θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που πιέζουν ε, η πολιτική μηχανή, ας πούμε, ατμομηχανή του προγράμματος αυτού, έτσι ώστε να γίνουν τελικά κάποια πράγματα στην, ε, στη βάση. Η βιομηχανική βάση σε κάποιες ε, χώρες είναι διαφορετική. Υπάρχει άλλες, σε άλλες χώρες μικρή, σε άλλες χώρες μεγάλη, ε, διαφορετική βέβαια για τον τομέα της άμυνας, αλλά πρέπει τα πράγματα να είναι σαφή. Να είναι σαφές δηλαδή ότι πάντα θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Ότι δηλαδή κάθε εθνική κυβέρνηση προφανώς πρώτα θα κοιτάξει τι έχει να αποφεληθεί η ίδια από τον τομέα της άμυνας. Αν τώρα μιλούμε για σημεία τα οποία βρίσκονται σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος όπου τελικά Μπορεί όντω η άμυνα μέσω τη δημιουργία θέσεων εργασία να δημιουργήσει ανάπτυξη στην περιοχή. Θα πρέπει ίσω να το, να το δούμε. Αλλιώ δεν έχει νόημα να δημιουργούμε δομέ. απλώς για να τις δημιουργούμε. Γιατί αν το δούμε μόνο ε, από την εθνική του πλευρά, θα, πρέπει, θα, θα χάσουμε ουσιαστικά την ευρωπαϊκή εικόνα και θα πρέπει να έχουμε μια γενική ευρωπαϊκή θεώρηση. Οπότε, το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε όλα αυτά, όλες αυτές τις σκέψεις που υπάρχουν ε, να τις συνδυάσουμε έτσι ώστε να προχωρήσουμε με τα αποτέλεσματα που θέλουμε σε όλους τους τομείς που θέλουμε να επιτύχουμε. Έχω υποβάλει κάποιες ε, ε, τροπολογίες γιατί στο, για, τον, για την πτυχή αυτή δεν είδα πολλά στο, στο κείμενο. Ε, η περιφερειακή ας πούμε, πολιτική, ε, σε αυτούς θα μπορούσαμε ίσως να απευθυνθούμε γιατί αυτοί έχουν κάποια κονδύλια. Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνεργαστούμε περισσότερο και με αυτούς, να ενισχύσουμε βέβαια τις περιφερειές τους προφανώς, αλλά και μέσω της συνεργασίας μας, ακριβώς επειδή ρέουν και άλλα κονδύλια σε αυτούς, να μπορέσουμε ίσως να έχουμε κάποια κοινά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της άμυνας ώστε να μην γίνονται αυτά μόνο σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές σε μια αγωνιά του πλανήτη. Και οι πολιτικοί λοιπόν και οι εθνικοί, των εθνικών κυβερνήσεων προφανώς έχουν κάποιο, ε, κάποια ανησυχία γιατί μπορεί να είναι αυτοί που τελικά θα χάσουν από όλη αυτή τη διαδικασία αν ας πούμε καταστραφεί ή καταρρεύσει μια τέτοια δομή. Αλλά η περιφερειακή πολιτική, ας πούμε, που παίρνουν χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία, ίσως θα μπορούσαν να είναι καλοί συνομιλητές με εμά για να μπορέσουμε να βρούμε τελικά μια κοινή λύση για το τι θα κάνουμε και πώς θα μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειές μας στον τομέα της άμενας, έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό τα ελλείμματα που υπάρχουν στον οικονομικό τομέα να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να τα καλύψουμε. Ευχαριστώ. Merci, euh, Madame Ευχαριστώ κύριε Νικολάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λίζα για την ε, μεγάλη και φιλόδοξη έκθεση. Έκθεση η οποία πιστεύω ότι καλύπτει πολλά θέματα. Οι οι στάσεις που διατυπώνει είναι πολύ σημαντικές. Θα ήθελα να παρατηρήσω το εξή. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι το ε, κάτι καινούριο στο πλαίσιο της κρίσης αυτής. Σίγουρα πλήτεται και από τη συγκεκριμένη κρίση η αμυντική βιομηχανία, αλλά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στον τομέα αυτό εδώ και πολύ καιρό, πολύ περισσότερο καιρό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε να βρούμε μια λύση ώστε την κρίση αυτή πράγματι να την κάνουμε ευκαιρία και πρέπει να επαναξιολογήσουμε όλες τις αμυντικές προτεραιότητες. Δυστυχώ δεν υπήρχε μακρά παράδοση συνεργασίας, είναι καιρός όμως τώρα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούμε στον τομέα της άμυνας. Ένα θέμα αυτό. Τώρα, βλέποντα την κοινή προσέγγιση, βλέπω ότι στην ιστορία μας είχαμε πολύ καλή συνεργασία, θυμάμαι το πολύ παλαιό αυτό πρόγραμμα Eurofighter που όμως ήταν μία από τις βέλτιστες πρακτικές συνεργασίας ή ένα άλλο ε, γαλλοϊταλικό πολύ επιτυχημένο σχέδιο στον τομέα του ναυτικού. Πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία αυτή, γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά κράτη-μέλη που έχουν κάποιες σκέψεις και κάποια οράματα σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες. Δεν συζητήσαμε σχεδόν καθόλου το θέμα της ε, διαλειτουργικότητας και αυτό πρέπει να συζητηθεί. Μπορεί να έχουμε τις δυνατότητες ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε ή να απαντήσουμε σε κάποιες απειλές, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και τη διαλειτουργικότητα των αμυντικών συστημάτων. Αυτό είναι πιο φθηνό. Είναι καλύτερο να υπάρχει η στενή συνεργασία λοιπόν και να ενθαρρύνουμε αυτή τη διασυνορική συνεργασία όπως την αποκαλούμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις συμβάσεις, τις προμήθειες για αμυντικό εξοπλισμό και εκεί θα πρέπει να έχουμε ένα κώδικα διοντολογίας. Θέλουμε να υπάρχει διαφάνεια και ανταγωνισμός ε, στην αμυντική βιομηχανία. Κάποιες χώρες το επιθυμούν, κάποιες άλλες όμως όχι. Δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενθουσιασμό προς αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει όμως να πιέσουμε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να προσχωρήσουν σε αυτή την προσπάθεια για να αποφύγουμε τη διαφθορά στο σύστημα των προμηθειών ε, για αμυντικό εξοπλισμό. Μπορεί να μην το συζητάμε, αλλά δυστυχώς υπάρχει πολλή διαφθορά στον τομέα αυτό. Έχουμε και τον ε, στόχο του Ελσίνκη για τον ε, κατάλογο ε, των δυνάμεων και δεν έχουμε την αξιολόγηση αυτού του project που παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει και θα πρέπει να μπορέσει να φέρει σε πέρα στις αποστολές Πέτερσμπουργκ. Είχαμε και στο Λάκεν τους στόχους που τέθησαν μέχρι το 2010. Σε ό,τι αφορά τώρα ε, την... Ε, of ε, την χωροφυλακή, κάτι πρέπει επίσης να σκεφτούμε. Πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες και να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση όλων των απειλών. Η χωροφυλακή ξέρουμε ότι συμμετείχε σε πολλές κοινέ πράξεις και δράσεις επιχειρήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Χωροφυλακής, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται και αυτή και να αντιδράσει. Στην ε, Σύνοδο Κορυφής Λισαβόνας είχαμε και την στρατηγική κυβερνοάμυνας. Έχουμε του χρόνου ε, το σχετικό πρόγραμμα για τις προμήθειες θα πρέπει να εφαρμοστεί. Είναι ένα νέο εμπόριο, ένας νέος τομέας και θα πρέπει κάπως να αντιδράσουμε. Θα πρότεινα με τροπολογίες μας ε, να συστήσουμε στα κράτη-μέλη να εξετάσουν ε, πολύ προσεκτικά αυτό το νέο είδος εμπορικών συναλλαγών και να δουν ε, τι δυνατότητες και παμπύλες θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Σε ό,τι αφορά την αγορά τώρα αμυντικού εξοπλισμού, σας πρέπει και αυτό να το συζητήσουμε, γιατί δυστυχώς δεν το έχουμε συζητήσει ουσιαστικά στο Κοινοβούλιο το θέμα των offset. Θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε και τη νομική υποστήριξη, αυτή την πτυχή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές καλές πρακτικές και υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία συνεργάζονται στην αμυντική βιομηχανία μέσω του offset. αμυντικές δυνάμεις ε, αγγλικές κτλ. Μία από τις βασικές προτεραιότητες που έχουμε είναι να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό, να μην φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να εξυγχρονιστεί και να έχει κοινά και ανταγωνιστικά σχέδια. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις και στην Εύρενα θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες όλων των κρατών μελών για να προωθήσουμε την έρευνα, διότι όλοι έχουν να προσφέρουν ε, ε, τη συμβολή τους στον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας, και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Έχουμε κάποιες προτάσεις, θα συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις. Δεν θα σας εκθέσω όλες τις τροπολογίες που θέλουν να καταθέσουν οι φιλελεύθεροι αυτή τη στιγμή, αλλά οφείλω να πω ότι η έκθεση είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι έχουμε την ευκαιρία ως Επιτροπή, ως Υποεπιτροπή, να δημιουργήσουμε νέες τάσεις και να δρομολογήσουμε εκ νέου τη συζήτηση για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε Κοπά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η διεθνή χρηματοοικονομική κρίση ε, δημιουργεί περιορισμού σε αμυντικές δαπάνε, αλλά ανακαλύπτει και κάποιες επίμονες αδυναμίες, οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατεπηγόντω. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Λίζεκ, γιατί είναι πολύ επίκαιρη η έκθεσή του δεν υπάρχει πραγματική επιλογή έναντι της μουσουλμικής πειθαρχίας. Όλοι το παραδεχόμαστε. Είναι αυτό αληθές για τα περισσότερα, αν όχι για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όπως ε, ήδη αναγνώρισαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, πρέπει αυτήν την κρίση να την δούμε ως ευκαιρία, όχι ως αδιέξοδο. Και θα πρέπει να τη δούμε ως ευκαιρία να έχουμε και να εφαρμόσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να επενδύσουμε με πιο σοφό τρόπο του πόρου μα και να αντιμετωπίσουμε σοβαρότερα την ε, ανάγκη καταπολέμηση τη διαφθορά ε, ε, στην όλη αγορά. Θα πρέπει να δούμε το pooling and sharing, την διοικητική μέρημνα και βέβαια να ενώσουμε τι προσπάθειε μα στον τομέα τη έρευνα και τη καινοτομία. Αυτή είναι η πρώτη συζήτηση, πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θέλω λοιπόν πέντε σημεία γενικού χαρακτήρα να αναφέρω αναφέρω και νομίζω ότι θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να επισέλθουμε σε περισσότερε λεπτομέρειε στην επόμενη συζήτηση. πρώτη παρατήρηση σε σχέση με την έκθεση. Πρέπει η συζήτηση να επικεντρωθεί περισσότερο στο πλαίσιο τη ΕΠΑ, να αναφέρουμε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλεια, η οποία ορίζει ε, και εντοπίζει τι απλέ και τι προκλήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τομέα τη άμυνα. Οι αμυντικέ ανάγκε καθορίζονται πράγματι από τι απειλέ, και πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να είμαστε ένα παράγοντα αξιόπιστο στο διεθνέ προσκήνιο και να τοποκριθούμε επιτυχώ, ε, ε, ιδίω εντό τη στενότερη περιοχή και θα πρέπει να ζητήσουμε την περιοχή και αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ε, Ασφάλειας και να ορίσουμε κοινού ε, στόχου, χωρί όμω να παραγνωρίζουμε τη χρηματοοικονομική κρίση. Πρέπει να ενώσουμε τι δυνάμει μα επομένω και να χρησιμοποιήσουμε του περιορισμένου πόρου που έχουμε στη διάθεσή μα με τον τρόπο που θα μας επιτρέψει να είμαστε ως τον πιο αποδοτικοί. Δεύτερη παρατήρηση, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα ποιοτικά μέσα όλες οι απειλές, ούτε πρέπει να ξεχνάμε το όφελος που θα είχε παγκοσμίω ε, η μη διάδοση όπλων και ο αφοπλισμός. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια παράδοση για τα μη στρατιωτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτο σημείο πρόταση αναδιαμόρφωσης ε, των ευρωπαϊκών βιομηχανιών με ανησυχεί, γιατί προτείνεται η επιλογή της συγκέντρωσης ε, και αυτό ε, θα δημιουργήσει δυσκολίες στο θέμα της απασχόλησης. Και έχουμε και την παράγραφο 37. Αν αυτή η αναδιάρθρωση αποτελεί αναγκαιότητα ή κάτι το αναπόφευκτο, θα πρέπει να τη δούμε ως μια ευκαιρία για να εδραιώσουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση, να δημιουργήσουμε νέες θέσει εργασία ενδεχομένω και να ανταποκριθούμε στο αυξανόμενο κόστο των αμυντικών εξοπλισμών και να εξασφαλίσουμε ε, την ασφάλεια του εφοδιασμού τέτοιο αμυντικού εξοπλισμό. Πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση, πρέπει να υπάρχει συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Αυτό σε συνδυασμό ε, με την ε, έκλεισε να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να ε, μειωθούν οι ελλείψεις και οι αδυναμίες που δημιουργούν προβλήματα στη βιομηχανική συνεργασία και βλάπτουν και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Τέταρτο σημείο. Συμφωνώ πλήρως ότι θα πρέπει να στηρίξουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και σε σχέση με το συντονισμό και το σχεδιασμό κοινών αμυντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Θα ήθελα ωστόσο να υπάρχει ευρύτερη συμμετοχή στα κοινά έργα και να υπογραμμίσω ότι επί, επί της αρχής, ως θέμα αρχής μάλλον, δεν θα πρέπει να αποκλείται κανένα κράτος μέλος. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει ε, μια διαδικασία που δεν θα διέπεται από την βιομηχανία, αλλά θα ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Και έρχομαι στο τελευταίο μου σημείο. Έχουμε διάφορε περιφερειακές πρωτοβουλίε pooling and sharing. Είναι καλή αρχή, τι ε, επικροτώ. Θα ήθελα όμω να ζητήσω να ληφθούν ε, περαιτέρω μέτρα και να υπάρξει πραγματική συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα θετικό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην έκθεση είναι η πρόσφατη απόφαση Ιταλία ή Ισπανίας να μπουν στην πρωτοβουλία τη. Ε, Βαϊμάρης. Βαϊμάρ. πρέπει να είναι ο κοινό μα στόχο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσκα για μια ακόμη φορά που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια προ, παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και την επόμενη φορά θα σας δώσω πολύ περισσότερες ε, λεπτομέρειες σχολιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συμφωνήσω και εγώ με όσους λένε ότι όντως είναι πολύ ε, κατανοητή και ενδιαφέρουσα η έκθεση του κ. Λίζεκ. πρέπει την οικονομική κρίση να την κάνουμε πλεονέκτημα και να δούμε πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να προωθήσουμε τι ιδέε τη κοινή άμυνα και τη ασφάλεια και τη σχετική πολιτική. Να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου Ράινχαρτ Μπούτικοφ γιατί δεν μπορούσε να είναι παρόν σήμερα. Οπότε ήθελα να σας αναφέρω εγώ αυτά που θα είχε να πει ο ίδιος ειδικά σε ό,τι αφορά την, ε, τις παραγράφους 29-32, με τις οποίες σχετικά διαφωνούμε, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μια συμβαστική λύση. Εγώ θα ήθελα, πέραν των όσων σχολείων ήδη ακούστηκαν, για την πολιτική άμυνας και ασφάλειας, να σχολιάσω και την συνεργασία της αερομαντικής βιομηχανίας. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία και νομίζω ότι αναφέρεται σωστά στην έκθεση, είναι το θέμα των κανονισμών και των κανόνων γενικώ για τους διαγωνισμούς. Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία όπου η βιομηχανία άμυνα ε, μπορεί να υποφεληθεί. Και η υπηρεσία άμυνα επίση είναι μια πολύ σημαντική, ε, έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πολλέ από τι ευρωπαϊκέ βιομηχανίε ανταγωνίζονται όχι μόνο στην εσωτερική αγορά, αλλά και στι εξαγωγέ του και θα ήθελα να ακούσω από τον κύριο Λίζεκ ποια είναι τα σχόλιά του για το σημείο αυτό και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Να διαχειριστούμε δηλαδή αυτόν τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Ε, ας πούμε η δημιουργία ενός κονσόρτσιουμ ή η αναδιάρθρωση είναι η μοναδική λύση. Ένα άλλο σχόλιο που έχω είναι η διεθνοποίηση της Ευρωπαϊκής Άμυνα, ε, Βιομηχανίας Άμυνας ποιος είναι ο ρόλος της στο, τώρα και στο μέλλον και πώς μπορούμε να, να αντιμετωπίσουμε αυτή την ε, ξένη ιδιοκτησία που όλο και περισσότερο αυξάνεται στον τομέα της άμυνας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούζινγκ. Ja, vielen Dank. Ευχαριστώ με πολλέ από τι παρατηρήσει ε, ε, και πολλών από του ε, συναδέλφου, κυρίω τη κυρία Κοπά, θα ήθελα να συμφωνήσω. Θα ήθελα όμω να ενισχύσω και κάποια πόσα ακούστηκαν. Προ το παρόν βρισκόμαστε σε μια πολύ αντικρουόμενη, αντιφατική κατάσταση. Η πρώτη αντίφαση, κατά δική μου άποψη, είναι ότι ευτυχώς έχουμε πολύ περισσότερη ειρήνη πλέον στην Ευρώπη, αλλά γεγονός είναι ότι η επικράτειά μας δεν ε, την χάνει επιθέσεων από πουθενά. Σε αντίθεση βέβαια με αυτό, έχουμε συνέχεια υψηλότερες δαπάνες για εξοπλισμούς και περισσότερες στρατιωτικές παρεμβάσεις εκτός Ευρώπης βέβαια. Και αυτό είναι βασικό για το θέμα που συζητούμε δηλαδή οι πολύ ε, λίγοι πόροι που υπάρχουν με τις, ε, σε σχέση με τις πολύ υψηλές ανάγκες που προκύπτουν από την στρατιωτική πλευρά, από τον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών. Η επόμενη αντίφαση, την είπανε και όλα οι συνάδελφοι, η ε, οικονομική, τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν από τα κράτη-μέλη. Και αυτό προκύπτει από την περιπλοκότητα του τομέα της άμυνας. Το είπε και η κυρία Κοπά, το είπαν και άλλοι. Πρέπει να θέσουμε το ερώτημα ποιος ορίζει τελικά τις δαπάνες για τον εξοπλισμό. Η βιομηχανία, η στρατιωτική βιομηχανία, τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών μελών ή όλα αυτά είναι απλώς κάποια απειλητικά σενάρια που έρχονται. Στη δική μου τη χώρα ε, έχει περάσει μια νομοθεσία που λέει ότι η Γερμανική, ο γερμανικός στρατός είναι καθαρά στρατός άμυνας. Και εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη που προέκυψε αυτό και θα ήθελα να πω σαφώς ότι οι απειλές ε, είναι απειλές σε μια επικράτεια. Μια ακόμη ε, αντίφαση που βλέπω βρίσκεται μεταξύ των δαπανών, των ε, ε, αξιοπλισμών και των δημοσιονομικών ε, προβλημάτων που αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη και τις περικοπές που πρέπει να κάνουν. Και θα ήθελα εδώ να πω ότι ας πούμε στην Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν συνάψει, έχουν πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να συνάψει συμφωνίες πολλών, ε, πολλών εκατομμυρίων για εξοπλισμούς. Η Ελλάδα έχει τους περισσότερους ίσως εξοπλισμούς σε όλη την ε, Ευρώπη. Παρόλα αυτά πρέπει ταυτόχρονα να κάνει και δραματικές περικοπές. Επίσης, άλλη αντίφαση μεταξύ των ευρωπαϊκών αξιών των αξιών δηλαδή της, ε, κοινό, της ευρωπαϊκής κοινότητας και της βοήθεια σε ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές κρίσεις. Υπάρχει και μια σχετική, υπάρχουν κάποια σχετικά πορίσματα τα οποία λένε ότι θα πρέπει να, ο αφοπλισμός να ε, παραμένει μόνο στο απόλυτο, στο ελάχιστο που χρειάζεται για να υπάρξει η απαραίτητη άμυνα για την κάθε επικράτεια. Για την, για την έκθεσή μου λοιπόν αυτή θα υποβάλω αρκετέ ε, τροπολογίε, γιατί σε κάποια από τα σημεία τη είμαστε τελείω διαφορετική άποψη. Ευχαριστώ. Merci. Ε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλαμ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η εκκίνηση που έκανε ο κύριος Λύση για να αντιμετωπιστεί μια δραματική κατάσταση. Μία από τις λέξεις κλειδιά της έκθεσης κατέμε είναι οι περικοπές άνευ προηγουμένου στις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες. Αυτό σημαίνει ότι θα υπονομευθεί η αξιοπιστία των αμυντικών μας δυνατοτήτων. Οι πόροι μας, τα μέσα μας ε, θα συνεχίσουν ε, να περιορίζονται και να προσπαθούμε να τα εκμεταλλευτούμε ώστε να τον περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τρεις ταυτόχρονες ε, κρίσεις. Δεν θα μπορούμε. Η Ευρώπη βέβαια πρέπει να, ε, και αν θέλει βέβαια, πρέπει πάντως να ε, πρωταγωνιστήσει και στο μέλλον, στο παγκόσμιο προσκήνιο. Και έχουμε τις συλλογικέ αμυντικές δαπάνες των 27 που αντιστοιχούν όπως και στο 1 τρίτο μόνο των αμυντικών δαπανών των ΗΠΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά βασικά προβλήματα τα οποία έχει επισημάνει ο συνάδελφος Λίζεκ. Ένα από αυτά είναι το pooling and sharing, αυτή η συγκέντρωση και κοινή χρήση δυναμικού. Αυτό πρέπει να θεωρηθεί αναγκαιότητα ε, και όχι πλέον επιλογή. Αν αυτό ισχύει, τότε ο ρόλο τη έρευνα και τη τεχνολογία, τις αμυντικές δαπάνε, αν περιορίζονται αυτέ στο 1% μόνο των συνολικών δαπανών, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ λίγος, δραματικά λίγος θα έλεγα. Και βέβαια η τυποποίηση του εξοπλισμού. Ουσιαστικά θα οδηγήσει στο να ξεπεραστούν τα εθνικά συμφέροντα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αν θέλουμε να διατηρήσουμε την αξιοπιστία μας και τη σοβαρότητά μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Πρέπει αυτούς τους εθνικούς διαχωρισμούς να τους ξεπεράσουμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε το δυναμικό των αμυντικών βιομηχανών και να το αξιοποιήσουμε. Τέλος, υπόθηκε ότι η χρηματοοικονομική κρίση είναι και μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να επιτύχουμε πρόοδο. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι αυτό πρέπει να φροντίσουμε να μην παραμείνει ένα σλόγγαν. Χρειάζονται σοβαρές προσπάθειες για να υλοποιηθεί. Περιμένω λοιπόν να εγκριθεί η έκθεση αυτή and uh, ώστε να εκπέμψουμε ένα ε, διακομματικό ισχυρό μήνυμα από πλευράς Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βέβαια και προς τα κράτη-μέλη. Προσβλέπουμε λοιπόν κύριε Λίζεκ στην επιτυχή έκβαση της έκθεσής σας. Ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστώ. Τελευταίος ο ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λίζεκ για το έργο που έχει επιτελέσει, που είναι πάρα πολύ αναλυτικό και πάρα πολύ σοβαρό. Εκπροσωπεί δε, από μάλλον, μια εξαιρετική αφετηρία για κοινή δουλειά μεταξύ των πολιτικών ομάδων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή αυτή. Θα ήθελα να αναφέρω δύο ε, σημεία πολιτικού χαρακτήρα, τα οποία ήδη προανέφερε η κυρία Κοπά. Εμείς ε, εκ μέρους της σοσιαλιστικής ομάδας θα θέλαμε να υπάρξει εμβάθυνση σε αυτά τα δύο σημεία. Ουσιαστικά δεν θα αναφέρουμε συγκεκριμένες προτάσεις ε, με τι οποίε είμαστε σύμφωνοι, θεωρούμε ότι είναι πολύ καλέ, αλλά αυτό το οποίο μα ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώ όλα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η αμυντική βιομηχανία μπορούμε να τα εντάξουμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο εν μέσω αυτής της χρηματοοικονομικής κρίσης. Πρόκειται για αλληλένδετα μεταξύ τους σημεία. Πρώτο, νομίζω ότι στην έκθεση αυτή πρέπει να γίνει μια επιλογή μεταξύ δύο πολύ διαφορετικών μηνυμάτων. Πρώτο μήνυμα είναι ότι η Ευρώπη δαπανά πολύ λίγα γιατί 200 δις είναι το 1 τρίτο μόνο των αμυντικών δαπανών των Και το δεύτερο μήνυμα είναι αφού δεν προβλέπεται να δαπανηθούν με περισσότεροι πόροι, και επειδή θα είναι μάλιστα και αναπόφευκτο να υπάρξουν μειώσεις, περικοπές, θα πρέπει να προβούμε σε πιο ευφυείς ε, δαπάνες, να δαπανούμε τα χρήματα που έχουμε με πιο ευφυή και με διαφορετικό τρόπο. Και θα πρέπει βέβαια να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τις δυνατότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα 200 δις ε, ουσιαστικά είναι το άθροισμα των 27 ε, εθνικών αμυντικών προπολογισμών. Και τι πετυχαίνουμε αυτά τα χρήματα, πετυχαίνουμε ε, τα ίδια πράγματα, μήπως υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις, άρα θα πρέπει να δούμε ε, το λόγο, τη σχέση μεταξύ πόρων και αποτελεσμάτων, που είναι μάλλον αρνητική η αναλογία θα έλεγα. Επομένως πρέπει να δούμε την ε, πτυχή της ευέλτιστης αξιοποίησης ε, των ε, δαπανών. Φυσικά και είμαστε υπέρ της ενίσχυσης των δυνατοτήτων του αμυντικού τομέα. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρούμε ότι επί του παρόντος η Ευρώπη δεν μπορεί καν να διανοηθεί αύξηση των αμυντικών δαπανών. Άλλο πρόβλημα. Είναι πολύ καλές και ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Πρόταση για ενίσχυση του pooling and sharing, συγκέντρωσης και κοινή χρήσης και πάρα πολύ ωραία λόγια όλα αυτά. Τι θα πει όμως συγκέντρωση και κοινή χρήση. Ουσιαστικά αυτή η έννοια περικλεί πάρα πολλές διαφορετικές έννοιες και θα πρέπει να εξεταστούν στην έκθεση αυτές οι πτυχές ε, από πολλά διαφορετικά πρίσματα μηχανισμός των Αθηνών, έρευνα, καινοτομία, τεχνολογία. Συμφωνώ, επαναλαμβάνω, με τις προτάσεις, αλλά κατά την άποψή μου οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν στη βελτίωση του ευρωπαϊκού αμυντικού τομέα. Τότε θα είναι Καλέ αυτέ οι προτάσει. αν δηλαδή μας δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια πραγματικά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνα. Τώρα πώ θα την αποκαλούμε, με ποια αρχικά, αυτό δεν με απασχολεί τόσο. Με απασχολεί το να είναι ευρωπαϊκή, πραγματικά ευρωπαϊκή αυτή η πολιτική. Στην έκθεση αυτή λοιπόν δεν πρόκειται απλά να αναφέρουμε και να επαναλάβουμε κάποια ισχυρά πολιτικά, θεσμικά επιχειρήματα κτλ. Συμφωνώ, πρέπει να είναι συγκεκριμένη η έκθεση, δεν είναι μια έκθεση η οποία αναφέρεται στο πολιτικό πλαίσιο γενικά και όπου ε, παραλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε το πνεύμα της έκθεσης, δηλαδή να υπάρξει μια στενότερη σχέση μεταξύ των προτάσεων που διατυπώνονται και της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Πάντοτε προς την προοπτική προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής. Πρόκειται για ισχυρές δεσμεύσεις. Θέλουμε να υπάρξει αλλαγή θεώρησης, αλλαγή νοοτροπίας και μια πραγματική κοινή χρήση των πόρων. Σίγουρα ε, υπάρχουν τα κεκτημένα, υπάρχουν οι κυριαρχίες εθνικές. Αν δεν ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική, η ευρωπαϊκή διάσταση, δεν θα μπορούμε να επιτύχουμε Μιλάμε για τον εξευρωπαϊσμό, αν θέλετε, της ε, πολιτικής άμυνας. Έχουμε δύσκολη δουλειά αν έχουμε να υπολογίσουμε για τις 27 διαφορετικές διαδικασίες σε επίπεδο δηλαδή κάθε κράτους μέλους. Η έκθεση είναι εξαιρετική πάντως ε, και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Λίζα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή για να καταλήξει. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αγαπητοί συνάδελφοι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους συντονιστές και όλους τους κοιόδες εισηγητές για τις παρατηρήσεις τους. Πάρα πολύ πολύτιμες όλες αυτές οι παρατηρήσεις. Άκουσα πολλές προτάσεις επικοδομητικές, για τις οποίες ε, χαίρομαι, και ε, ενστάσεις ή ερωτηματικά ε, με ικανοποίηση που μου τα θέσατε, αλλά σήμερα δεν μπορώ να απαντήσω. Αν είχα τις απαντήσεις άλλωστε, ξέρετε, σε όλα αυτά τα ερωτήματα, μάλλον θα είχα μια, ένα πολύ υψηλότερο αξίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα ζητήματα αφορούσε τον ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός ουσιαστικά είναι και ο λόγος για τον οποίο αντιμετωπίζουν προβλήματα πολλές χώρες και πολλά εργοστάσια ευρωπαϊκά. Θυμάμαι όταν συνομιλούσαμε κάποιον ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τον τομέα της άμυνας, Είχε μάλιστα διατελέσει υπουργό Άμυνα στη χώρα του και τώρα έχει μια σημαντική θέση πάντα σε αυτόν τον τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συγκεκριμένο αυτό άτομο μου είχε πει. Ε, μα πώς ε, εσείς περιμένετε να έχετε αποτελεσματικά εργοστάσια ε, στην Ευρώπη. Αν θέλουμε στην ε, Ευρώπη να έχουμε τέσσερα διαφορετικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ στη ΣΥΠΑ έχουν δύο εργοστάσια και παράγουν έναν μόνο τύπο τέτοιου αεροσκάφους. Πώς θέλετε να είναι αποτελεσματικά τα εργοστάσια τα ευρωπαϊκά, όταν επίσης δημιουργείται και θέμα με τις εξαγωγές. Δεν μπορούν να εξαγάγουν. Έχουμε 16 εργοστάσια στην Ευρώπη επίσης τα οποία ε, κατασκευάζουν ε, άρματα μάχης τεθωρακισμένα. Στις ΕΠΑ τρία είναι αυτά τα εργοστάσια. Και οι ευρωπαϊκές ανάγκες είναι πολύ χαμηλότερες σε σχέση με τις αμερικανικές ανάγκες. Το ίδιο ισχύει και με τα ε, αεροσκάφη. Ή έχουμε επίσης πολλά ναυπηγεία τα οποία ναυπηγούν ε, πολεμικά πλοία. Και αντίστοιχη κατάσταση παρατηρούμε αν συγκρίνουμε τη ΣΥΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είναι ατυχής η κατάσταση και είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα αυτών των εργοστασίων. Είναι πολλά εργοστάσια αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα να πουλήσουν και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Επίσης αναφέρατε πάρα πολύ σημαντικές πτυχές πολιτικού χαρακτήρα. Πολύ εξ αναφέρατε το θέμα της συνεργασίας. Είπατε μάλιστα ότι πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς, όχι μόνο τους υπουργούς άμυνας βέβαια, αλλά και στις, ε, στα Εθνικά Κοινοβούλια ή στις Επιτροπές Άμυνας των Εθνικών Κοινοβουλίων των Κρατών Μελών. Ο κύριος Γκάλερ μίλησε για την πολιτική συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί στο περιφερειακό επίπεδο οι πολιτικοί έχουν έναν όλο και σημαντικότερο λόγο σε ό,τι αφορά τη βιομηχανία και τη βιομηχανική παραγωγή των χωρών τους. Πολλοί επίσης με ρώτησαν ε, για το ποιος είναι ο βασικός αποδέκτης αυτής της έκθεσης. Ουσιαστικά ε, ξαναθέσατε με τις ερωτήσεις σας αυτό το, το ζήτημα, δηλαδή τι εξυπηρετεί αυτή η έκθεση, σε τι θα ωφελήσει. δεν είναι μόνο το να έχουμε ε, την εντύπωση ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Ο στόχος μας είναι να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα σε όλους τους ε, πολιτικούς σε κάθε επίπεδο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ε, συνεργασία και σίγουρα θα μπορέσουμε να εκπονήσουμε μια έκθεση η οποία θα έχει ένα ισχυρό μήνυμα και η οποία θα τύχει υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόκειται για μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, για τις προθεσμίες, για τις τροπολογίες 19 Οκτωβρίου. Και θα τις εξετάσουμε στις 10 Νοεμβρίου. Ένα μήνα έχουμε μπροστά μας, ο Κριστόφ ε, Λίζεκ ε, διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές ομάδες. Στείλτε λοιπόν όλες σας τις τροπολογίες και παρατηρήσεις αυτές τις εβδομάδες. Προχωράμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Καλό τον Αλέν Ρουά να έρθει στο βήμα.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε με το δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τον ε, κύριο Λερουά, ο οποίος έφυγε, ε, εγκατέλειψε το, τη θέση του ως αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ και πρώην διευθυντής ε, του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων για να τα πω σύντομα δηλαδή των ε, κοιονοκράνων. Έχει μακρά εμπειρία ε, στην ε, διαχείριση των σειράξεων και των μεταπολεμικών καταστάσεων. Ε, ήταν κατά τον πόλεμο στο Σεράγεβο 94-95 μετά ήτανε αναπληρωτής ε, γενικός ε, γραμματέας. Ε, θα λέγαμε ότι ε, αρμόδιος για το Κόσοβο, θα λέγαμε ένα είδος νομάρχη. Μετά πήγε στην πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όπου βοήθησε για την έξοδο από την κρίση το 2001. Ήσασταν και πρεσβευτής της Γαλλίας στη Μαδαγασκάρη. Είστε εξοικειωμένος δηλαδή με τις ρηψοκίνδυνες περιοχές. Οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΟΗΕ είναι μια πολύ έντονη ανησυχία της Επιτροπής μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των κρίσεων. Θέλω λοιπόν να σας ακούσω, να μας πείτε πώς βιώσατε εσείς ως Ευρωπαίος αυτή την εμπειρία σας στον ΝΟΙΕ. Ενδιαφερόμαστε επίσης από την θεσμική σας εμπειρία. Θέλουμε να μας πείτε περισσότερα δηλαδή για το τμήμα ειρηνευτικών επιχειρήσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς λοιπόν να σας ακούσουμε. Κυρίως αυτά που έχετε να μας πείτε για την Αφρική, που αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο ανάπτυξης ειρηνευτικών επεμβάσεων στην ακτή του Ελεφαντόδοντος παίξατε έναν ε, σημαντικότατο ρόλο, βοηθήσατε και στη γέννηση ενός νέου κράτους του Νοτίου Σουδάνα, Πολλές λοιπόν αφρικανικές ε, ε, ε, πολλά γύρω από την αφρικανική επικαιρότητα. Τώρα εσείς πλέον δεν είστε, δεν έχετε, δεν έχετε επίσημα το αξίωμα, άρα έχετε και μεγαλύτερη ελευθερία λόγου. Τώρα δίνω και το λόγο στον Αντιπρόεδρο Πάσκου γιατί συνδιοργανώνουμε με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Να σας καλωσορίσω και εγώ εκ μέρους της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, έχετε τεχνική κατάρτιση, ξέρετε λοιπόν ε, πολλά, έχετε εμπειρία από την θεσμική σας θέση και στη Γαλλία και στις εξωτερικές σχέσεις στον ΟΗΕ, οπότε πραγματικά είσαστε ένα μεγάλο μια, μια πηγή πλούτου γνώσεων και εμπειριών. Οπότε παρακαλώ έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Υποεπιτροπής Ασφάλειας, ε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι βούλευτες, θα μιλήσω εγώ ως πρώην γενικός ε, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Εχθές ε, ορκίστηκε ο διάδοχός μου. Θα σας αναφέρω λοιπόν πολύ ε, σύντομα ε, για το ιστορικό πλαίσιο, θα σας αναφέρω και διδάγματα από ορισμένε περιπτώσεις, Σουδάν, Κονγκό, ακτή του Ελεφαντόδοντο, λίγα για το Αφγανιστάν, και τρίτο για τις δράσεις που χρειαζόμαστε σήμερα για να μπορέσουμε να ανασυνταχθούμε. Και να πω επίσης τι θεωρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πράττει σήμερα, πώς θα μπορούσε να πράξει περισσότερα. Πολύ σύντομα να θυμίσω το τι σημαίνει διατήρηση της ειρήνης. 120.000 στρατιώτες, 180 συνολικά μεταξύ στρατιωτών, αστυνομικών και πολιτικού προσωπικού, 22.000. Δηλαδή μετά από τον Αμερικανικό στρατό πρόκειται για, αυτό το ένα δις ε, δολάρια είναι ένας προϋπολογισμός ε, αντι, αντίστοιχος με τον Ηνωμένων ε, με τον προπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς πέρυσι, είμαστε, πριν από 10 χρόνια ήμασταν 20.000 και δέστε που φτάσαμε. Το 2011 είχαμε δύο νέες επιχειρήσεις για τον, στο Σουδάν για το Νότιο Σουδάν και για το hot spot μεταξύ νο, Νότου και Βορρά. Και αυτό για να μπορέσουμε να απαντήσουμε γρήγορα στις και έγκαιρα στις κρίσεις. Να σας θυμίσω ότι το 48 ξεκίνησαν οι πρώτες ειρηνευτικές διαδικασίες, ακόμη και αν δεν το είχαμε στη χάρτα του ΟΗΕ, είναι η NSO στη Μέση Ανατολή, ένσω. Υπάρχει ακόμα ως δράση, παραδοσιακές δηλαδή δράσεις για τη διατήρηση της ειρήνης αυτή, στο Κασμίρ το 49 που συνεχίζει να υφίσταται στην Κύπρο, τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το 64, 800 δηλαδή άνθρωποι που συνεχίζουν να παρακολουθούν την ε, διαχωριστική γραμμή και μετά έχουμε την Έντορφ στον Κολάν που και εκεί πάλι πρόκειται για παρατήρηση. Από, δηλαδή μπαίνουμε ανάμεσα στους ε, Σύριους και στους ε, Ισραηλινούς που κατέχουν το Γκολάν. Αυτό είναι το παραδοσιακό μας, το κλασικό μας πλαίσιο. Βέβαια οι ειρηνευτικές πλέον παρεμβάσεις δεν έχουν πλέον αυτόν τον χαρακτήρα, είναι ευρύτερε και πιο πολυδιάστατες για το Κονγκό. Στην ε, ε, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ε, η εντολή του ΟΙΕ καλύπτει 41 διαφορετικές αρμοδιότητες να βοηθήσουμε τον στρατό κατά των επαναστών, να βοηθήσουμε για τις εκλογές, να μεταρρυθμίσουμε τον τομέα της ασφάλειας, ε, ε, βοήθεια για την ολοκλήρωση κλπ. Βλέπετε δηλαδή σήμερα οι δράσεις μας είναι πολύ πιο ευρείες, πολύ πιο πολιτικές, άρα και πιο πολύπλοκες. Μερικά για τις νέες προκλήσεις αυτών των επιχειρήσεων στις οποίες η Ευρώπη μπορεί να συνεισφέρει ιδιαίτερα. Να υπογραμμίσω ότι έχουμε τρία νέα ζητήματα. Πρώτο, η πολυδιάσταση, ο αριθμός των αρμοδιοτήτων, των καθηκόντων που έχουμε. Τρίτο, ο οπλισμός που είναι πολύ πιο βαρύς, διότι πρώτα εμείς χρησιμοποιούσαμε τα όπλα μας για αυτοάμυνα αλλά πλέον τα χρησιμοποιούμε και για την προστασία της εντολής. Το κάναμε στην ακτή του Λεφαντόδοντος αλλά και στο Κονγκό. Είχαμε ας πούμε επιθετικά ελικόπτερα στο Κονγκό τα οποία πυροβόλησαν κατά των επαναστατών σε δύσκολες περιπτώσεις. Πάντοτε δηλαδή και ανόκρανη, αλλά σε πιο σκληρές ε, καταστάσεις. Η πολιτική εμπειρία, ε, μπορεί η ευρωπαϊκή εμπειρία μπορεί να μας βοηθήσει στην προστασία των, του αμάχου πληθυσμού. Και έχουμε μία πρόταση στην εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας που λέει μέσα σε μία πρόταση και μόνο, πολύ εύκολη πρόταση, ε, δηλαδή προστασία του αμάχου πληθυσμού, απλούστατη πρόταση, αλλά πολύ δύσκολη ε, να υλοποιηθεί στον ε, επιτόπου. Η προστασία του αμάχου πληθυσμού είναι μια δουλειά ιδιαίτερα σημαντική, δύσκολη και διαφορετική από το να πολεμάει κανείς που είναι πράγμα για το οποίο είναι προετοιμασμένοι οι στρατιώτες μας. Και γύρω από αυτό έχουμε σε συνεργασία με εσάς αναπτύξει νέες στρατηγικές. Φυσικά στο Κονγκό έχουμε δολοφονίες, έχουμε βιασμούς ε, γυναικών παρά το γεγονός ότι είμαστε παρόντες. Έχουμε δηλαδή ακόμη πολλά να κάνουμε, αλλά βέβαια προχωρήσαμε στα τελευταία χρόνια, βελτιωθήκαμε. Διδάγματα για πρόσφατες ε, κρίσεις και σχόλια για τις πρόσφατες κρίσεις. Για το Σουδάν. Ε, ε στο Σουδάν έχουμε πράγματα τα οποία ε, έγιναν πολύ σωστά. Αρχές Ιανουαρίου, 2 Ιανουαρίου του 2011 το δημοψήφισμα πήγε πολύ καλά και έχουμε και αλλού δυσκολίες και μου λέγανε ε, οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι ότι ούτε καν το φανταζόντουσαν ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό το δημοψήφισμα και καλά και χωρίς βία. Και καμιά δεκαπενταριά αρχηγοί κρατών εμφανίστηκαν τον Μάρτιο στον για όταν συζητούσαμε το θέμα του Σουδάν και κατάφεραν να πιέσουν τη Χαρτούμ να κρατήσει τις προθεσμίες. Αλλά για την περίπτωση του Σουδάν η αμερικανική πολιτική πίεση ήταν πολύ πιο σημαντική από ότι η ευρωπαϊκή πίεση. Εγώ ως Ευρωπαίος θα ήθελα να υπάρχει μια μεγαλύτερη πολιτική εμπλοκή της Ένωσης ε, στο Σουδάν. Ε, εγώ έλεγα πριν από χρόνια στο ΚΑΠΣ, ΚΟΠΣ, ότι το Σουδάν είναι πολύ σημαντική χώρα. Η αστάθεια του Σουδάν θα δημιουργούσε αστάθεια σε όλη την Αφρική. Είναι μια χώρα που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη. Και μετά είχαμε τον ε, κύριο Τόμπεν Μπρίλ και την, μετά την κυρία Μάτσεν ε, ως αντιπροσώπους εκεί, αλλά δεν είχαμε μεγάλη παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, αλλά σας το λέω έτσι για να προσπληροφόρηση. Να τελειώσω με το Σουδάν. Η κατάσταση δεν είναι απόλυτα ρυθμισμένη. Είναι οι 193 ε, χώρα των, του ΟΗΕ. Βέβαια τα πράγματα ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί. Πρόκειται για μια τεράστια χώρα. Ε, έχουμε 7.000 Γάλλους στρατιώτες εκεί. Αλλά ξέρετε ότι οι σχέσεις στις παραμεθόριες περιοχές μεταξύ ε, βορρά νότου μέχρι τις μέχρι τον Κιανούν Νίλο ε, έχουμε μεγάλα προβλήματα και θα έπρεπε να έχουμε πιέσεις και προς τη Ζούμπα και προς το Χαρτούμ. Δηλαδή δίνονται μάχες και έχουμε νεκρούς ε, κάθε, κάθε χρόνο. κάθε μέρα, συγγνώμη. Και στον Ταρφούρ η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ δύσκολη. Έχουμε δύο εκατομμύρια εκτοπισμένους ε, στο Ταρφούρ. Είναι μια χώρα η οποία απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους της Ευρώπης. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό πρόκειται για μια τεράστια χώρα όπως όλοι γνωρίζετε. Πρόκειται για μια χώρα η οποία δεν μπορεί να δικήσει την επικράτεια και ο ΙΕ είναι παρόν εκεί από το 1960. Θα θυμάστε την, τον θάνατο του Ντάγλες Μάρσελ ε, ε, στο Κονγκό. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν κάνει τεράστιες προόδους τα τελευταία 5-10 χρόνια. Δεν έχουμε πλέον αλλοδαπούς στρατούς στο Κονγκό. Η κατάσταση έχει σχετικά ηρεμήσει. Αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε εκλογές. Οι όροι ε, κάπου πληρούνται για να μπορέσουμε να, έχουμε αυτές τις εκλογές. Το Βέλ... Έγινε μια τεράστια προσπάθεια, το Βέλιο μας δάνεισε ένα 630, έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες ε, από την Ευρώπη και από τότε που απειλήθηκε η γκόμα ε, στα ανατολικά από τις ΕΝΤΕΠΕ, όταν είχα αναλάβει εγώ μάλιστα τα καθήκοντά μου, είχα επισημάνει ότι θα έπρεπε να φανταστούμε ένα ευρωπαϊκό μάχη μοτάρ με ένα battle group, αλλά μου απάντησαν, μου απάντησαν όχι. Ευτυχώς όμως η κατάσταση τελικά σταθεροποιήθηκε. Ακτή του Λεφαντόδοντος, άλλη περίπτωση. Όλοι σας γνωρίζετε τι συνέβη γιατί τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα. Συνολικά η κατάσταση σήμερα στην ακτή του Λεφαντόδοντος έχει κάπως σταθεροποιηθεί. Έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, ο πρόεδρος που εκλέγει θα αναλάβει την εξουσία, είχαμε νεκρούς σε μετεκλογικές ε, συγκρούσεις, υπάρχει μια διεθνής επιτροπή για να δει ποιο είναι ο υπεύθυνο. Ο, κύριος, ο πρόεδρος Γουατάρα είπε ότι εντάξει θα ήθελε να αποδοθεί δικαιοσύνη. Εκεί εμείς ε, είχαμε αποφασίσει να πλήξουμε τους ε, στόχους που ήταν βαριά όπλα που έπληταν, που ε, χτυπούσαν τον πληθυσμό. Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτά τα βαρέα όπλα ήταν βαρέα όπλα του Προέδρου Μπαγκμπό και στις 4 Απριλίου αυτό όταν έδωσα τη διαταγή να χρησιμοποιήσουμε τα όπλα μας Βέβαια ήξερα πάρα πολύ καλά ότι είχα κοντά, ήταν κοντά οι ειδικέ δυνάμεις Λικόρν της Γαλλίας και, μπορούσαν να αποτελέσουν ενίσχυση, είχαμε ενισχύσεις δηλαδή για μία εβδομάδα για μία εβδομάδα τρεις μέρες κράτησε. Και αυτό ήταν ένα πραγματικό δίδαγμα αυτό το οποίο συνέβη για να συνειδητοποιήσουμε τις ανάγκες μας για τη Λιβύη. Ξέρετε ότι στη Λιβύη, δεν έχουμε peacekeeping. Πρόκειται για μια επέμβαση του ΝΑΤΟ με εντολή του ΟΗΕ και ο κύριος ανασμούσεν κάθε φορά που συναντάει τον Μπανκιμούν του λέει ότι τα πάντα βρίσκονται υπό την εντολή του ΟΗΕ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ εξέφρασε τη βούληση να είναι πάντοτε υπό την εντολή του ΟΗΕ. Δεν έχουμε λοιπόν peacekeeping. Υπάρχει όμως μία πολιτική αποστολή του ΟΗΕ έτοιμοι για τη βοήθεια στο, στη σύνταξη του συντάγματος, στην κατάρτιση της αστυνομίας, στην οργάνωση εκλογών κλπ. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν αυτό το, αυτή την... Ε, έχουμε προετοιμάσει αυτή την αποστολή, η οποία δεν είναι αποστολή peacekeeping, αλλά είναι αποστολή για την επίβλεψη αν διατηρείται η κατάπαυση του πυρός. Αν δηλαδή θα υπήρχε κατάπαυση του πυρός και έπρεπε να επιβλέψουμε ότι θα διατηρηθεί ή όχι. Ξέρετε όμως ότι τα πράγματα δεν πήγαν έτσι. Πήγαν αλλιώς, κάπως έτσι πήγαμε. Τώρα έχουμε την πολιτική αποστολή, την ΦΙΑΣΛ στο Αφγανιστάν που έπαιξε σημαντικό ρόλο στις εκλογές και στη συντήρηση του κράτους δικαίου. Μπορώ να απαντήσω μετά στις ερωτήσεις σας βέβαια για το καθένα από αυτά τα θέματα. <clears throat> Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 10, 15 δράσεις σήμερα. Συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε 64 τέτοιες δράσεις, 45 έχουν κλείσει. Έχουμε 15 δηλαδή σήμερα που παραμένουν από την Αϊτή στο Τιμόρ, μέσω Κωσυφοπεδίου, Λιβερίας κλπ. Δεν μιλάμε πια για αυτά, αλλά όσοι ενδιαφέρονται, ας πούμε στη Λιβυρία τα πράγματα αλλάξανε και θα έχουμε εκλογές. Ε, στο Τιμόρ επίσης ε, ε, τα πράγματα πάνε καλά, ελπίζουμε να κλείσουμε την αποστολή και το ότι Μοριανό συγγραφέα βραβείο Νόμπελ και θα έρθει στον ΟΗΕ να μιλήσει για αυτά. Πάντως τέλος πάντων διαπιστώνεται ότι όπου πάμε εμείς επιφέρουμε σταθερότητα, σχετική σταθερότητα στις χώρες που επισκεπτόμαστε. Πέρυσι. Και στο παρελθόν. Τι έγινε. Είχαμε πετυχημένες δράσεις. 2003. Άρτεμις, ανατολικά του Κονγκό, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έστησε μία δράση για δύο-τρεις μήνες, όπου ναι μεν εμείς πηγαίναμε για peacekeeping, αλλά δεν είχαμε τον οπλισμό και τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε να αντιμετωπίσουμε τους επαναστάτες. Εγώ πήγα στον Ιτούρι πριν από 6 μήνε και στον Ιτούρι πάνω από 600 άτομα, 6 ε, ε, εκατομμύρια συγγνώμη, άτομα έχουν επιστρέψει στα σπίτια του. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση της Ένωσης αυτή ε, η δράση Άρτεμις. Επίσης, η ΕΦΟΡ το 2006 στο Κονγκό πάλι όπου επιτράπηκαν έτσι οι πρώτες εκλογές συνολικά σε όλη την επικράτεια. Πραγματικές δημοκρατικές εκλογές στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και αυτό με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν υπήρχε δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις εκλογές. Άλλη δράση πιο πρόσφατη. Εφόρ στο Τσάντ. Ξέρετε ότι με το, από τον Ταρφούρ οι πρόσφυγες πήγανε στο Τσάντ, πολύ δύσκολη κατάσταση ανατολικά, στο ανατολικό Τσάντ και, το, και ο ΙΕ ήταν αρκετά αργός να αναπτύξει τις δυνάμεις του. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρώπη μετά από πολλές και αποφασιστικές συζητήσεις αποφάσισε να στείλει για ένα χρόνο το 2008, 15 Μαρτίου με 15 Μαρτίου, ε, να στείλει στρατεύματα στο Τσάντ. Και το 2009 εγώ ήμουνα στην ε, Τζαμένα όπου έγινε η ανταλλαγή των πηλικίων όπου οι Ευρωπαίοι στρατιώτες αντάλλαξαν τα πηλίκια με αυτούς του ΟΙΕ. Βέβαια, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν θέλει να δεσμεύεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ε, γι' αυτό δεσμευτήκανε για ένα χρόνο στο Τσάντ, γιατί ο ΙΕ μετά μπορεί να δεσμευτεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτά είναι για παράδειγμα, βέβαια τα πάντα δεν είναι τέλεια. Ο συντονισμός ε, δεν ήταν ιδιαίτερα, ε, δεν ήταν ιδιαίτερα προβληματικός, είχαμε και προβλήματα με τη χρηματοδότηση. Τώρα, <clears throat> το ανάποδο, Κωσυφοπέδιο. Το Νοέμβριο του 2000, α, τον 9 Δεκεμβρίου του 2008, διορθώνεται ο μιλητής. Ε, περάσαμε εμείς τις αρμοδιότητες, περάσαμε την εξουσία στην ΕΛΕΞ, ε, δηλαδή την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν απόλυτα λογικό δηλαδή να αναλάβει τα ενία η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εκεί βρισκόμαστε μέσα σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και στο Κωσίφο και στη Σερβία. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη στα σύνορα. Αλλά η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε πολύ σωστά. Υπάρχουν και άλλοι τομείς γύρω από τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ε, Πολ και σε δύο αποστολές της Ένωσης στο Κονγκό. Ας πούμε έχουμε μετρικά δελτία για τον κάθε στρατιώτη, τα οποία μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε στρατιώτης πληρώνεται. Επίσης η ΕΠΟΛ στο Αφγανιστάν για την κατάρτιση της αστυνομίας. Βέβαια 400 αστυνομικοί ή χωροφύλακες βρίσκονται εκεί. Ο αριθμός, ε, έχουν συγγνώμη καταρτιστεί, ο αριθμός αυτός δεν είναι τόσο σημαντικός, αλλά αν ξέρει κανείς την κατάσταση εκεί, ε, ε, ήδη καλά είμαστε με αυτόν τον αριθμό. Στην ΑΕΤ τώρα. Στην IT μας είπανε θέλουμε χωροφύλακες και τους είπαμε εμείς θα στείλουμε τους Ευρωπαίους χωροφύλακες στην Γαλλική Ζανταρμερή, τους Ιταλούς καραμπινιέρους αλλά δεν οργανωθήκανε και δεν πήγανε. Έχουμε μετά την Αταλάντα, την άλλη δράση την οποία σας ευγνωμονούμε. διότι οι ευρωπαϊκές νιοπομπές βοηθάνε ιδιαίτερα στην καταπολέμηση της πειρατείας στη Σομαλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης καταρτίζει τους, τους, ε, <laughs> τους στρατιώτες της προσωρινής ε, κυβέρνησης της ε, Σομαλίας. Υπάρχει όμως μία τεράστια μια διαφορά, μια τεράστια διαφορά μεταξύ των επενδύσεων για την Αταλάντα 500 ε, εκατομμύρια δολάρια ή δεν ξέρω τι και την προσπάθεια on shore Ξέρουμε ότι οι λόγοι της πειρατείας, οι αιτίε της πειρατείας είναι on shore Θα έπρεπε τα συνέπεια να καταρτήσουμε σωμαλούς, αστυνόμους και στρατιωτικούς ε, για να υπάρξει μικρότερη δυσαναλογία μεταξύ της επένδυσης που γίνεται offshore και της προσπάθειας που καταβάλλεται onshore. Για να ολοκληρώνω τρεις τομείς για τους οποίους θα μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία της με τον ΟΗΕ. Οι προϋπολογισμοί άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται. οι δράσεις του ΟΗΕ συνήθως πάνε εκεί που κανένας άλλος δεν θέλει να πάει, η Λιβερία ή η Κονγκό. Θα παραμένει δηλαδή απαραίτητη αυτή η παρέμβαση διατήρηση της ειρήνης. Η Ευρώπη στηριοποιηθεί σε άλλους τομείς. Συμμετοχή. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν πολύ σημαντική το 1990. στη χρηματοδότηση του peacekeeping ήταν η μεγαλύτερη καθαρός εισφέρουσα. Το Πακιστάν, Ινδία και το Μπαγκλαντές είναι οι μεγαλύτεροι χορηγοί σε στρατεύματα. Μετά έχουμε την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και μετά την Αυστρία. Αλλά η Αυστρία είναι ο 400 συνεισφέρον σε στρατεύματα. Συνολικά οι ευρωπαϊκές δυνάμεις μεταξύ των 120 είναι 6.900 6.900 στρατιώτες. Μιλάω για τους ένστολους, οπότε πρέπει να υπολογίσουμε καμιά κατοσταριά χιλιάδες. Σε αυτές τις 100.000 έχουμε 6.900 Ευρωπαίους, και 5.400 είναι στο Λίβανο, στη Φινούλ. Μεγάλη επιχείρηση. Οι Ιταλοί, Γάλλοι, οι Ισπανοί και άλλοι Ευρωπαίοι, Φιλανδοί, Δανέζοι κλπ. που αλληλοδιαδέχονται ένα στον άλλον. Ένα κόμμα δηλαδή στην συνεισφορά ενστόλων. Πρέπει ακόμη να καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. όταν ξέρουμε δηλαδή ποια είναι και η τεράστια επένδυση της Κομισιόν στα διάφορα αναπτυξιακά σχέδια στην Αφρική. Θα μπορούσατε λοιπόν να κάνετε παραπάνω, 1,7 είπαμε, η συμμετοχή. Οι ευρωπαϊκές χώρες επίσης χρηματοδοτούν το 40% των διαφόρων επιχειρήσεων. Τεράστια ανισορροπία δηλαδή μεταξύ χρηματοδότησης και στρατευμάτων. Δεύτερο, εξοπλισμός μιλούσα για την βαρύτητα των διαφόρων επιχειρήσεων. Ε, σίγουρα έχουμε τον εξοπλισμό που χρειαζόμαστε στο Λίβανο, αλλά θα χρειαζόμασταν και αλλού. Τα αεροπλάνα, τα νυχνευτικά αεροπλάνα ντρόν, χωρίς πιλότο. Μέγα μέρος του στρατού μας δεν τα έχει αυτά τα αεροπλάνα. Επίσης έχουμε αυτά τα περίφημα ελικόπτερα και ελικόπτερα ε, μεταφορά στρατευμάτων αλλά και ε, μαχητικά ελικόπτερα, έχουμε πολιτικά ελικόπτερα, τα νοικιάζουμε, εύκολο είναι, αλλά δε, λόγω ε, συνθήκων συμβολέων και ασφαλείας και λοιπά δεν μπορούμε εμείς να πάμε σε επικίνδυνες περιοχές διότι τα συμβόλαια μας τα απαγορεύουν με τα νοικιασμένα. Άμα αποσυρθούν βέβαια τα, άμα πάρετε πίσω τα ελικόπτερά σας από το Κονγκό καήκαμε. Επίσης αυτή η αντίληψη, αυτή η ιδέα των στρατευμάτων over the horizon, πέρα του ορίζοντος, σε περίπτωση κρίσης χρειαζόμαστε ενισχύσεις πολύ συγκεκριμένες, σε συγκεκριμένους τομείς. Θα μπορούσε η Ευρώπη να μας βοηθήσει. Τέσσερις-πέντε περιπτώσεις είχαμε τα τελευταία χρόνια. Ανέφερα το Κονγκό, Εφόρ και Άρτεμις, αλλά Σιέρα Λεόνε, δέστε. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε πάρα πολύ, για, για, για πάρα πολύ λίγο να μας βοηθήσει να σταθεροποιήσουμε τη χώρα και τελειώσαμε. Πλέον εκεί δεν έχουμε ανοιχτή επιχείρηση, δεν έχουμε ανοιχτή δράση, έχει σταθεροποιηθεί η χώρα. Άλλο παράδειγμα, ΑΕΤ μετά από το σεισμό του Ιανουαρίου 2010. Για τέσσερις μήνες ήρθαν οι 20.000 Αμερικανοί στρατιώτες που δεν ήταν πολύ μακριά, ήρθαν να βοηθήσουν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν ήρθαν με καμιά δεκαριά ε, πλοία και 20.000 στρατιώτες για να μας βοηθήσουν. Και για την ε, Λικόρν ε, στην ακτή του Ελεφαντόδοντος και εκεί είχαμε μια πολύ σύντομη επιχείρηση. Αυτή είναι η συνεισφορά που μπορώ να φανταστώ για τα ευρωπαϊκά κράτη. Και μετά αυτή η αντίληψη του Battle Group που, άμα, που βλέποντάς το δηλαδή με το μάτι του ΟΗΕ, του Τμήματος Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων, ε, Αυτό είναι, αυτό θα ήταν ιδιαίτερα καλό. Βέβαια παραμένει ακόμα ανοιχτό η Ευρωπαϊκή χώρα να το δεχτεί και μετά να τον εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτά τα battle group θα ήταν πολύ χρήσιμα. Στο chat είχαμε μιλήσει και σε κάποια φάση για τα battle group, αλλά αυτό δεν, τελικά δεν ήταν η λύση που υπερίσχυσε. Και για το Κονκότα το προτείναμε, μας είπαν όχι. Καταλαβαίνω ότι για τη Λιβύη ένα μέρος το οποίο χρησιμοποιείται ε, και πιο συγκεκριμένα από τις Σουηδικές δυνάμεις ε, ε, θα μπορούσαν να αποτελούν κομμάτι των Battle Group, δεν έχουν όμως ακόμα χρησιμοποιηθεί επίσημα. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξετάσουμε και αυτό το μέσο των Battle Group. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά... Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να είστε σύντομοι και συγκεκριμένοι όταν λαμβάνετε το λόγο. Από πλευρά μου τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο στο οποίο εργάζεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Έχετε κάποιες ειδικέ διευθετήσεις και, και κανονισμούς ε, κατά περίπτωση ή ένα πιο διαρθρωμένο, πιο δομημένο διάλογο. Ποιοι είναι οι συνομιλητές σας στην προκειμένη περίπτωση. Με ποιον ε, μιλάτε, με τον ύπατο εκπρόσωπο, με την ύπατο στην προκειμένη περίπτωση, με τον επικεφαλή της ΚΟΠΣ και δεύτερον, η σχέση σας με την Αφρικανική Ένωση, ιδίως ε, αν δούμε και την περίπτωση της Ομαλίας, δύο χώρες ουσιαστικά συνεισφέρουν, Μπουρούντι και Ουγκάντα. Έχουμε συναντηθεί πολλοί από μας με εκπροσώπους των δύο χωρών αυτών και παραπονούνται σε ό,τι αφορά ε, την παραγωγή δυνάμεων, αν θέλετε, για τη χώρα αυτή. Και τελευταίο, πιο προσωπικό ερώτημα, σε σχέση με την ευρωπαϊκή εμπειρία που έχετε. Υπήρξατε δικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στα Σκόπια, με εξωτερικό μάτι και ως ε, τέος ευρωπαϊκός πάλι εντό εισαγωγικών, πώς εσείς βλέπετε ε, την ε, ίδρυση της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχετε κάποια σχόλια. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάμσντορφ, ε, που είναι επικεφαλής της ομάδας μελετών Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Εθνών, όπως γνωρίζετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα Α, να το κάνω στα αγγλικά ίσως είναι πιο εύκολο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την παρέμβασή σας. Είμαστε μαζί στην αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στη Νέα Υόρκη και κάποια από τα ερωτήματα που θα έθετα εγώ μόλις τα έθεσε ο Πρόεδρος, οπότε θα είμαι πάρα πολύ σύντομος ειδικά σε ό,τι αφορά την αλλαγή του, της ε, Γενικής Γραμματείας, του interface, δηλαδή από τη Γενική Γραμματεία στην Υπηρεσία Εξωτερικών Σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη δική σας την δουλειά. Πώς έχει επηρεάσει τη δουλειά σας και αν έχει βελτιωθεί η δουλειά σας με την αλλαγή αυτή. Επίσης, άκουσα να μας ζητάτε να επηρεάσουμε περισσότερο την, ε, τις ε, υπηρεσίες στην Αφρική, γιατί οι περισσότερες από τις ε, παρεμβάσεις που μας αναφέρατε βρίσκονται στην Αφρική. Υπάρχει ένα πρόβλημα βέβαια, το οποίο είναι ταυτόχρονα και, ε, και ευκαιρία, γιατί είναι το απικιακό ας πούμε παρελθόν των κρατών μελών. στο Κογκό ας πούμε είχατε βελγικά ελικόπτερα, στην Αχτή του Λεφαντοστού είχατε γαλλικά ελικόπτερα. Ε, υπάρχει περίπτωση σε αυτή την μεταπικιακή ε, συμπεριφορά των, των κρατών μελών να αλλάξει κάτι, γιατί είναι προφανώς ε, πολύ διαφορετική, πολύ δυσανάλογη η προσοχή που λαμβάνουν κάποια κράτη, κάποια κράτη της Αφρικής από κάποια, σε σχέση με κάποια άλλα. Κάποια δηλαδή δεν τη χάνουν καμίας προσοχή. Αυτά. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήταν ε, πάρα πολύ σύντομο, συγκεκριμένο και σαφές. Εμπνευστείτε οι υπόλοιποι. Κυρία Κοπά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λερουά. Θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη και θα επικεντρωθώ σε μια συγκεκριμένη πτυχή της παρουσίας των κιανοκράνων. Για χρόνια, και ιδίω ό,τι αφορά την Αφρική, υπήρξαν πολλές καταγγελίες για συμμετοχή των κιανοκράτων σε βιοπραγίες και συγκεκριμένα σε βιασμούς. Έχετε μιλήσει γι' αυτό ε, και σήμερα μιλήσατε γι' αυτό, αλλά γενικά εγώ δεν άκουσα εκ μέρους σας μια σοβαρή αυτοκριτική για τον τρόπο στρατολόγησης των ε, κιανοκράνων, ιδίως αυτών που προέρχονται από γειτονικέ χώρες ε, της Αφρικής, ούτε αυτοκριτική για το σύστημα που άφησε λίγο πολύ ανεξέλιγκτη την παρουσία των κιανοκράνων στα διάφορα μέρη της Αφρικής. Εγώ ε, ακούω να επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα χωρίς να αλλάζει τίποτα όμως. Πάντως ε, διονίζονται αυτά τα φαινόμενα, οι βιοπραγίες και οι βιασμοί. Μπορεί να αλλάζουν τα ονόματα, αλλά παραμένει το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να μου δώσετε μια πιο ξεκάθαρη απάντηση, γιατί είναι ένα θέμα πραγματικά ανθρωπιστικό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λέζινγκ, έχει τώρα το λόγο. vielen Dank. Ευχαριστώ. Πολλοί οι τομεί που αναφέρθηκαν, πολλά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα απλώ να επικεντρωθώ σε δύο πραγματάκια. Μιλήσατε για την ε, εντολή, η οποία πρέπει να είναι πιο ισχυρή κάθε φορά. Και είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε αυτοάμυνα και θέλετε, λέτε, πιο ισχυρές και πιο συγκεκριμένες ε, εντολές. Νομίζω ότι θα έπρεπε εδώ να πούμε ότι αυτές αυτή η εντολή ουσιαστικά είναι εντολή ε, από το κεφάλαιο 7 και όχι εντολή από το κεφα... που απορρέει από το κεφάλαιο 6. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να βασίζονται σε μια τελείως διαφορετική βάση. Γιατί υπάρχει εδώ και θέμα ποσοτικό. Γιατί το κεφαλαίο 6 και οι σχετικέ ε, εντολέ που απορρέουν από αυτό μιλά, μιλούν για ε, συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Ενώ στι υπόλοιπε εντολέ δεν συμβαίνει αυτό οι δικέ σα παρεμβάσει παρεμβάσεις και οι επιχειρήσεις για τις οποίες μιλήσατε, ας πούμε η εντολή του ΟΗΕ ε, για τη Λιβύη ή για την παρέμβαση στο νακτή του του, ουσιαστικά σημαίνει ενίσχυση ενός από τους εμπλεκόμενους στην ε, όλη σύραξη. Και στο τέλος μετατρέπονται οι, ε, οι στρατιωτικές μονάδες συνυπεύθυνους για την πολεμική κρίση που υπάρχει στην ε, κάστοτε χώρα. Οπότε, μήπως θα πρέπει να, στο μέλλον να γίνουν προσπάθειες μέσω διεθνούς δικαίου να τροποποιηθεί η κατάσταση αυτή, ώστε να αλλάζει αναπερίπτωση. Και επίσης, ένα ερώτημα για την ΑΕΤ. Την αναφέρατε. Και τις τελευταίες μέρες διάβασα ότι εκεί αρχίζουν και γίνονται, αρχίζει και υπάρχει μεγαλύτερη αντίσταση από τον πληθυσμό κατά τον, του στρατιωτικής μονάδας του ΟΗΕ. Ε, θα παρέμβετε εσείς σε αυτό. Τι θα κάνετε με την αντίσταση αυτή και πώς δικαιολογείτε η μεγαλύτερη ακόμα ε, παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεων σε μια τέτοια χώρα σε μια χώρα δηλαδή που δεν ε, επιθυμεί καθόλου την ύπαρξη των στρατιωτικών μονάδων του ΟΗΕ. Εσεί πώ ακριβώ το δικαιολογείτε, τι ε, συμπεράσματα βγάζετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λερουά. Να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν θα είμαι εδώ να ακούσω τις απαντήσεις σας, αλλά θα μου τα πει όλα ο βοηθός μου που θα παραμείνει. Δεν πρέπει να πάω σε μια λεπτοπή να ψηφίσω. Λοιπόν, ποια είναι τα ερωτήματά μου. Πρώτον, έθεσε η κυρία Κοπάη, συνάδελφός μου, ε, το θέμα των κριτηρίων ε, στρατολόγησης για το πώς θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε ε, αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττονται από στρατιώτες των Ηνωμένων Εθνών. Τι γίνεται σε επίπεδο προετοιμασίας Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι καταλαβαίνει ο κόσμος, καταλαβαίνει τα καθήκοντα που έχει να φέρει σε πέρας, ότι έχει την ευθύνη να προστατεύει το human security, αυτήν την έννοια. Το έχουν στο κεφάλι τους, το έχουν στο μυαλό τους στρατιώτες. Επόμενο ερώτημα. Οι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τα κράτη-μέλη μα, μεταξύ άλλων. Φαντάζομαι και από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα μου πείτε εσεί. Τι αντίκτυπο μπορούν να έχουν σε αυτή ακριβώς την έννοια ε, της δημιουργίας ευθύνης, το, το, καθήκον της προστασίας, προστασία ανθρωπινών δικαιωμάτων. Σημείωσα αυτό που είπατε και το ερώτημα του Προέδρου. Έχει η Άμισομ την εντολή που πρέπει να έχει. Μιλήσατε για τη Λιβύη και για ένα σχέδιο έκτακτη ανάγκη το οποίο έχετε σχεδιάσει. Όταν μιλάμε για την ασφάλεια των συνόρων, θα μπορούσε αυτό το πλαίσιο, αυτό το πρόγραμμα να το αξιοποιήσετε. Και επειδή υπάρχουν φόβοι από πλευρά ε, ε, των Λίβιων ότι μπορεί να υπάρξουν ε, απόπειρε αποσταθεροποίηση από γειτονικέ χώρε. Τέλος. Ψήφισμα 1325 για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε όλες τις επιχειρήσεις και στο τμήμα ερευνητικών επιχειρήσεων. Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα. Στη Λιβερία συγκεκριμένα νομίζω έχουμε ένα αστυνομικό σώμα το οποίο παρτίζεται από Ινδές γυναίκες αποκλειστικά. Θα μπορούσατε να μας δώσετε άλλα παραδείγματα που ε, δείχνουν και στα άλλα κράτη ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερες γυναίκες σε επιχειρήσει σε αποστολές και στο τμήμα των ερευνητικών επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ, αλλά έχει το λόγο. θα προσπαθήσω να είμαι και εγώ συγκεκριμένος και συνοπτικός. Το πλαίσιο των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι. Έχουμε τον διάλογο κατά εξάμεινο ε, με τους διάφορους φορείς και με τις υπηρεσίες της εκπροσώπου. Γενικός διάλογος αυτός ε, αλλά σε συνάρτηση ε, με την κάθε αποστολή ε, προσαρμοζόμαστε κάθε φορά στις απαιτήσει του διαλόγου. Ο διάδοχός μου τώρα θα είναι αρμόδιος για το διάλογο αυτό. Προσπαθούμε να τον κάνουμε πιο συγκεκριμένο το διάλογο με την ε, ναι, αυτή υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι δεν υπήρχε ικανοποίηση από το επίπεδο ρεαλισμού του διαλόγου αυτού και νομίζω ότι τώρα θα πρέπει, αντί να είναι γενικό ο διάλογο, να βάζουμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Λιβύη, Σουδάν, εξοπλισμό, αυτά τα ζητήματα πρέπει να τίθενται επιτάπητο. Και όχι κατά περίπτωση να συζητάμε. Ε, αυτό που θέλω να πω σε ό,τι αφορά την ΕΙΕΔ και εμείς βέβαια από το Τμήμα Μερευτικών Επιχειρήσεων εμείς είμαστε έτοιμοι, στην ΕΕ τώρα οργανώνονται, αλλά έχουμε τακτικές επαφές, η κυρία Άστον, ε, ε, με τους διάφορους managing directors ε, που χειρίζονται τους διάφορες υπήρους και σε ό,τι αφορά την Υπάρχουν επαφές, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει στον τομέα αυτό μια προσπάθεια βελτίωσης της διάτρωσης του διαλόγου μεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση με τις τελευταίες χρονιές. Είμαστε προσκολλημένοι στο ad hoc ε, επίπεδο, στο κατά περίπτωση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΕΕΔ και το πώς μπορώ να την αξιολογήσω, Δεν είναι... είχε, είχε υποθεί ότι για τη Γαλλική Επανάσταση είναι πολύ πρόσφατη για να μιλήσει κανείς, δεν θα πω το ίδιο. Είμαστε ακόμα πάντως σε μια φάση που έχουμε συνεχείς επαφές, σταθερές επαφές. Εγώ ήμουν κάθε έξι μήνες στο ΚΟΠΣ και το ίδιο θα κάνει και ο διάδοχός μου. Στι αντιπροσωπείε του κοινοβουλίου, είχε έρθει και είπατε εκπρόσωπο ε, ε, στη Νέα Υόρκη κάθε δύο-τρει μήνε. Την έβλεπα ή εγώ ή το managing director. Άρα έχουμε έναν ε, διάλογο Απλά νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πλήρως δομημένος από εδώ και πέρα αυτός ο διάλογος. Σίγουρα δεν είναι ξεκάθαρα ακριβώς ποιοι θα είναι οι ρόλοι του Managing Director, η MDP. Ε, από πλευράς Νέας Υόρκης δεν τα βλέπουμε πολύ ξεκάθαρα ακόμα. Ούτε και εμείς λέμε πρόεδρος. Λοιπόν, ε, εντάξει, ε, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα μπουν στη θέση τους όλα αυτά και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα πιο δομημένο διάλογο σε σχέση με μέχρι τώρα. Σχέσεις με την Αφρικανική Ένωση πολύ σημαντικός εταίρος για εμάς φυσικά. 60 με 70% των επιχειρήσεών μας είναι στην Αφρική. Και σε ό,τι αφορά την Άμισον, δηλαδή την επιχείρηση Σομαλία, πάρα πολύ λεπτή επιχείρηση, πολύ ευαίσθητη, γιατί στα τέλη του 2008 η κυβέρνηση Ιμπούς ήθελε να είναι ε, το Εθνών η επιχείρηση. Σομαλία είχα εγώ ε, αντισταθεί σε αυτό και πολλές χώρες ε, της Ευρώπης με υποστήριξαν δεν είναι peacekeeping, αλλά peace enforcement. Δεν υπήρχε ε, διατήρηση της ειρήνης, γιατί δεν υπήρχε ειρήνη. Έπρεπε να επιβληθεί, να εγκαθιδρυθεί η ειρήνη. Και έτσι είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή επιχείρηση, πάρα πολύ δαπανηρή και ε, το Μπουρούντι, η Ουγγάντα, στο Μογκαντήσου έκαναν σημαντική δουλειά. Έχασαν πολλούς άντρες όμως, έχασαν πολλούς στρατιώτες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η επιχείρηση αυτή. Δεν ήταν ειρηνευτική με την έτσι της διατήρησης ειρήνης, αλλά με την έτσι επιβολή της ειρήνης, επαναλαμβάνω. Ήταν peace enforcement και όχι peace keeping. Εμεί δεν μπορούσαμε να έχουμε τη συγκατάθεση των κρατών μελών μα για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια αποστολή. Η Ουγγάντα και το Μπουρούντι, επαναλαμβάνω, έκαναν καταπληκτική δουλειά. Το θέμα είναι, η Αφρική Ένωση ζητά rehatting, όπως λέγεται, ε, αυτή τη επιχείρηση, να γίνει δηλαδή ε, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Προσπαθούμε να το περάσουμε, αλλά νομίζουμε ότι ακόμη είναι λίγο νωρίς για να γίνει αυτό, διότι έχουμε ακόμη συγκρούσεις, έντονες συγκρούσεις ε, και έμψω στο Μογκαντήσου πάλι ε, λίγο εύθραυστη είναι ως αποστολή. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Τώρα, ο νέος πρέσβης επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη μας βοηθά πολύ ήταν ε, ο Αυστριακός ε, πρέσβης και ήταν και μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας για δύο χρόνια. Ξέρει πάρα πολύ καλά, συμμετείχε σε επιχειρήσεις μας, έχει οργανώσει πολλά σεμινάρια και στην Νέα και στην Αυστρία για το θέμα αυτό. Άρα ε, νομίζω ότι ο εκπρόσωπος αυτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΕ θα διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί γνωρίζει και τον ΟΗΕ και έρχεται από την ΕΕ. Θα ήταν πολύ σημαντική λοιπόν η συμβολή του πιστεύω για τον κύριο Λάμσντορφ. Η στάση των χωρών στην Αφρική. Επειδή κάποιες είναι πρώην επικοκρατικές δυνάμεις, έχουν μια ισχυρότερη βόληση να αναλάβουν δράση. Πράγματι, έτσι είναι τα πράγματα. Είπα ότι οι Βρετανοί πήγαν στη Σιέρα Λεόνε, οι Λικόρνε στην ακτή του Όλα αυτά είναι ξεκάθαρα, έτσι και στην εκπαίδευση κτλ. Στη Λιβυρία ή παντάξει, δεν είναι πρώην επιτοκρατική δύναμη, αλλά τέλο πάντων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα αυτή. Για μα χρήσιμο είναι αυτό, γιατί υπάρχουν χώρε που ενδιαφέρονται και άρα όταν προκύψει ανάγκη μπορούμε να επικαλεστούμε τη βοήθειά τη. Στο Βέλγιο για το Κονγκό, τελικών, ε, ε όπω σα είπα, ή ξέρω εγώ ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα που ενδιαφέρεται για μια χώρα της Αφρικής, αλλά θέλουμε να μετριαστεί ο ρόλος των πρώην απειτοκρατικών δυνάμεων, δηλαδή να παρεμβαίνουν ε, όχι σε διμερές πλαίσιο χώρες, αλλά σε ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο. Θα ήταν καλύτερο ε, και θα ήταν πιο αποδεκτό από τις διάφορες χώρες. Να υπάρχει δηλαδή μια ευρωπαϊκή και όχι μια διμερής απάντηση ενός ευρωπαϊκού, συγκεκριμένου ευρωπαϊκού κράτους. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε για την κυρία Κοπά τώρα, που μίλησε για κάτι διαφορετικό. Sexual exploitation and abuse το λέμε αυτό στην ε, ορολογία μας, ε, σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Λέτε ότι δεν αλλάζει τίποτα βέβαια, ε, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Πράγματι, ε, τα μίντια κάθε φορά που υπάρχει μια περίπτωση τέτοια, ένα κρούσμα στο Κονγκό, και στην Αιτή με ένα τρομερό από Ρουγουανού ε, στρατιώτες που επρεσάν σε βιασμούς εκεί. Ε, αυτά προβάλλουν τα μίντια, αλλά έχουν γίνει και θετικά, πολλά θετικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, διαφάνεια. Έχουμε εμεί στο σελίδα εδώ και δύο χρόνια, όπου απογράφουμε, καταγράφουμε κάθε ε, κρούσμα το οποίο έχει καταγραφεί για βιοπραγία από στρατιώτες του ΟΗΕ. Μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα αυτό, Business Security. Υπάρχει λοιπόν αυτή η προσπάθεια για διαφάνεια. Δεύτερον, απαιτούμε από τις χώρες να επιβάλλουν κυρώσεις στα άτομα τα οποία διαπράττουν τέτοιου είδους ε, ενέργειες. Υπάρχουν χώρες πιο διστακτικές από άλλες, αληθεύει αυτό, αλλά πολλές χώρες πλέον το κάνουν. Η Γαλλία όταν υπήρξε ε, νομίζω ήταν βιασμό ανήλικη ε, στο Κονγκό, ένας Γάλλος στρατιώτη, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια νομίζω κάθριξη. Ο Ουρουγουανός αυτός που σα είπα επίσης, ο πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ουρουγουάης, ε, ε, κάλεσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο της ΑΕΤΗΣ και έγινε δημόσια δίκη για το στρατιώτη αυτό. Έγινε μια, υπήρξε πολύ μεγάλη προσοχή και προβολή αυτή τη υπόθεση. Υπάρχει ε, μεγάλη προσπάθεια. Επίση, καταβάλουμε επίση προσπάθεια στον τομέα τη πρόληψη και τη εκπαίδευση. Δηλαδή, στη στρατολόγηση, όταν ε, έρχεται ένας νέος στρατιώτης, προσέχουμε να μην έχει κακό ιστορικό στον τομέα αυτό. Και επίσης ε, παρέχουμε εκπαίδευση στο pre-deployment training όπως το λέμε και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία ε, στον τομέα αυτό και είναι το οποίο όλες μας τις δυνάμεις επιμένουμε, λέμε ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοια πράγματα. Πρώτα απ' όλα για έναν στρατιώτη, αλλά ιδίως για έναν στρατιώτη που είναι σε μια ειρηνευτική αποστολή να διαπράττει τέτοιου είδους ε, εγκλήματα. Και έχουμε κινητοποιήσει όλους μας τους εκπαιδευτές. Και για να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό, θα το δείτε και στην ιστοσελίδα μας, ένα αριθμητικό στοιχείο θα σας δώσω μόνο. Ο αριθμός θυμάτων, πώς να το πω, καταδικών, καταγγελιών μάλλον, έχουν ε, μειωθεί σημαντικά. Ε, ήταν πάνω από 300 τα άτομα πριν από 5 χρόνια που ε, κατηγορούνταν, ενώ τώρα έχουμε 84 άτομα μόνο. Γι' αυτά υπάρχουν ε, ε έρευνες. Δηλαδή 84 κρούσματα σε 120.000, ξέρετε, το Abu Ghraib, ε, άμα συγκρίνουμε αυτά, δυστυχώς ε, υπάρχουν αυτά τα μελανά σημεία σε κάθε στρατό. Επαναλαμβάνω, 84 περιπτώσεις 120.000 και ανώκρανους. Βέβαια υπάρχουν και Πολιτική, μη στρατιωτικοί ε, αξιωματικοί οι κάνουν. Λοιπόν, εμείς προσπαθούμε με την πρόληψη, με τη διαφάνεια. Ο Μπάνκι Μούνο, Γενικός Γραμματέας, ε, επιμένει και εγώ όταν ήμουν ε, πρόεδρος, επίσης μονίμως ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Συνεχίζεται λοιπόν ξέρω να υπάρχει μεγάλη προβολή σε αυτά τα παράδεκτα φαινόμενα, αλλά έχει μειωθεί δραματικά, έχει μειωθεί εντυπωσιακά ο αριθμός τέτοιων περιπτώσεων. Κυρία Γκέζινγκ, για την εντολή πράγματι. Οι εντολές είναι όλο και πιο πολύ κεφαλαίο 7. Πολύ μεγαλύτερη ισχύς της εντολής. Ξέρετε την έκθεση Μπραχίμη του 2000 που έλεγε ότι δεν θα πρέπει να μένουν stand-by και ανόκρανοι για την περίπτωση που θα δεχθούν επίθεση ε, πολίτες φυσικά και πρέπει να είναι πιο ισχυρή, robust. Ε, και εξού εφαρμόστε όλο και πιο πολύ το κεφάλαιο 7. Το ερώτημά σας ήταν νόμιμο ή όχι, γιατί πράγματι βλέπουμε κάποιες φορές ε, να αντιμετωπίζονται οι στρατιώτες του ΟΗΕ ως ε, παράγοντες ενεργοί μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Στη Λιβύη, να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι μια επιχείρηση από την αιγίδα του ΟΗΕ, όχι όμως ειρηνευτική. Απλά υπάρχει εντολή που μπορεί να δώσει ο ίδιο, όποιον το επιθυμεί να παρέμβει. Όταν έχουμε λοιπόν μία επιχείρηση, αυτό γίνεται πάντοτε με τη συγκατάθεση των μερών. Όταν δεχθεί ο Γενικό Γραμματέα, δηλαδή, επιχείρηση peacekeeping, πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση. Είχαμε τώρα την περίπτωση τη εκτό του ελεφαντοστού, τότε είχαμε συγκατάθεση των μερών. Ένα όμω μέρο απέστρεψε την συγκατάθεσή του. Αυτό ήταν διαφορετικό. Δεν θα είχαμε στείλει ειρηνευτική αποστολή εάν ε, είχε αποσύρει, η τότε που απέσυρε τη συγκατάθεσή του ένα μέρος. Είχε εγκριθεί από πριν η αποστολή. Τώρα, για τη Λιβύη, είναι νόμιμο ή όχι. Εγώ ε, θα σα παραπέμψω στην χάρτα των ομεθνών που την έχουν υπογράψει όλα τα μέλη του, που λέει ξεκάθαρα το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει την ευθύνη, την πρώτα αρχική ευθύνη σε θέματα ειρηνή και ασφάλειας στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι όλες οι νομικέ υπηρεσίες αναγνωρίζουν ότι οι αποφάσει του Συμβουλίου Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών έχουν νομική ισχύ. Δεν το έχει αμφισβητήσει αυτό ποτέ κάποιο ε, νομικό τώρα. Κατά πόσον από πολιτική πλευρά είναι θεμητό ή όχι, αυτό είναι άλλο ερώτημα. Αλλά από νομική πλευρά νομίζω ότι ε, καλύπτεται από τη Χάρτα των Εθνών. Στην περίπτωση Τη Λιβύης έχουμε το ψήφισμα 1973 και κάποιοι είπαν ότι η ερμηνεία που έγινε ήταν πιο ε, ευρεία και την αφισβήτησαν. τέλο πάντων, το ψήφισμα το ίδιο ε, και η εντολή του ε, δεν νομίζω ότι έχει αμφισβητηθεί νομικά. Εξ όσων γνωρίζω. Τώρα το πώ υλοποιείται η εντολή αυτή, αυτό είναι άλλο. Αλλά η ίδια η εντολή, η νομιμότητα τη εντολή δεν έχει αφισβητηθεί από κανέναν. Και αν κάποιος θέλει να αφισβητήσει, μπορούσε να θέσει ε, το βέτο. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα για τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου ασφαλεία. Τώρα έρχομαι στην ΑΕΤ. Είπατε, και έχω και εγώ διαβάσει στον τύπο, να γίνεται λόγος για το ότι ένα μέρος του πληθυσμού είναι δυσαρεστημένο με τη δράση του ΟΗΕ επιτόπου. Το έλεγα και στον τύπο στην Νέα Υόρκη δυστυχώς, μάλλον δεν είχα πολύ επιτυχία, σε όλες τις δραστηριότητές μας βλέπουμε τον τύπο να επικεντρώνεται συγκεκριμένα και αποκλειστικά στο 5% ε, που δεν ε, ε, λειτουργεί σωστά, δηλαδή στο 5% των τρένων που καθυστερούν και όχι στο 95% που φτάνουν στην ώρα τους. Φυσικά και υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν ή δεν θέλουν να έχουν μια δύναμη κατοχή στη χώρα τους. Και το λένε και το γράφουν και στους στίχους. Και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν κατηγορήσει την Μινούστα ότι ε, έβαλε μέχρι, μέχρι και τη χολέρα στην αίτη. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποδείξει επιστημονικά βέβαια. υπάρχουν τέτοιες ε, κατηγορίες. Αλλά ο ε, πληθυσμός στην πλειοψηφία του είναι υπέρ της διατήρησης της μηνωστά στην IT. Είχαμε αυξήσει ε, κατά 2.000, σε 2.000 άτομα ε, τη δύναμη αυτή μετά το σεισμό θα τη μειώσουμε τώρα κάτω από τα 2.000 άτομα. Αλλά νομίζω ότι η πολιτική τάξη, ιδίω στην ΑΕΤ, καταλαβαίνει ότι αν φύγει η Μουστά τότε θα υπάρχει χάος και θα υπάρξει ε, μεγαλύτερη δυστυχία και πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στη χώρα. Εμείς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε και την αστυνομία της ΑΕΤΗΣ, αλλά ε, υπάρχουν τα ζητήματα κατά πολέμηση των συμμοριών, μετά είχαμε την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού και ο κύριος Μαρτέλη ήδη και άκουσε ένα μέρος του πληθυσμού να λέει ότι δεν θέλει ε, τη Μινουστά, αλλά ο ίδιο είπε ότι όχι, πρέπει να μείνει η δύναμη αυτή. Υπάρχει το χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση. Είπε ότι θα είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνο για τη χώρα να γίνει αυτό ε, απότομα. Σίγουρα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός, ίσως να είναι λιγότερο ορατή. Και έχουμε και αυτό την περίπτωση του Ουργουανού που σας είπα που ε, προέβησε βιασμό. Φυσικά και δεν ε, δικαιολογούνται όλα αυτά και όλα αυτά πρέπει να αποτραπούν. Είναι πρόωρη απόσταση από την ΑΕΤ όμω και δεν το θέλουν και οι ίδιες οι πολιτικές, η ε, ε, πολιτική τάξη της χώρας. Τι άλλο είχα να απαντήσω. Κριτήρια στρατολόγηση και εκπαίδευση. Από την κυρία Γκομές που ε, έπρεπε να φύγει. Ναι, πράγματι. Φυσικά και προτείνω όταν ξεκινάμε μια αποστολή, προτείνω σε όλες τις χώρες να συμμετάσχουν σε ό,τι αφορά τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα ε, των γυναικών και το human security. Φυσικά και μας ενδιαφέρει. Αναπτύσσουμε, όπως σας είπα, ε, τα θέματα αυτά, ε, δικαιώματα των γυναικών, ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση που κάνουμε. Φυσικά και δεν είμαστε ποτέ τέλειοι και εργαζόμαστε με χώρες που δεν είναι και τα καλύτερα παραδείγματα στον τομέα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εξού και ακόμη περισσότερο αναγκαίο να στραφούμε στις ευρωπαϊκές χώρες και να συνεργαστούν περισσότερο μαζί μα. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα περισσότερο. Περισσότερη συνεργασία με τι ευρωπαϊκέ χώρε. Σε ό,τι αφορά τι ιδιωτικέ εταιρείε ασφαλεία και τον αντίκτυπό του ε, στον ΟΗΕ είναι πολύ αμελητέ η ποσότητα. Μόνο στο Αφγανιστάν έχουμε ε, κάποιες, ε, κάποια μέρη και που προσ, τις προστατεύουν οι ιδιωτικές εταιρείε. Αλλιώς δεν μας αφορά και πολύ το θέμα αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που ετέθη όμως είναι η ευθύνη προστασίας μείζον θέμα. Να σας πω εμπαρόδο ότι αυτή η πρόταση στο ψήφισμα για τον κοινοτικό του του δεν είναι μέσα. Μόνο στη Λιβύη. Όχι στο 1973, αλλά και στο 1970. Εκεί για πρώτη φορά έχουμε αυτή την λέξη σε μελάν και χαρτί. Ήταν το κεφαλαίο 7, όπως είπε η κυρία πριν από τη Γερμανία, Η ευθύνη λοιπόν για προστασία είναι κάτι καινούριο που αναφέρεται. Εμείς έχουμε αυτή την ευθύνη, αλλά είναι και ένα λεπτό θέμα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στους τέσσερους τομείς που ψήφισαν το 2005, δηλαδή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου, γενοκτονίες και εθνοκάθαρση. Αυτά τα τέσσερα εγκλήματα είναι αυτά των οποίων το 2005 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισε, ενέκρινε αυτή την ευθύνη για προστασία. Υπάρχει λοιπόν ε, ολόκληρη συζήτηση ακόμη στο επίπεδο του ΟΗΕ σε σχέση με τους τέσσερις τομείς αυτούς. Προς το πάνω περιοριζόμαστε εκεί. Τώρα για τη Λιβύη επανέρχομαι. Οι αναλυτές θα το κρίνουν βέβαια, κατά πόσον ε, εφαρμόστηκε σωστά και το ψήφισμα 1970 και το 1973. Δεν μπορούμε να πούμε αν πραγματικά ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σωστά αυτή η ευθύνη για προστασία. Ένα άλλο ερώτημα για την άμυσα στη Σομαλία από την κυρία Γκόμε πάλι. Υπήρχαν πράγματι μέχρι τώρα 8.000, τώρα θα γίνουν 12.000. Και στην Αφρικανική Ένωση μας λένε συνέχεια θέλουμε 20.000, χρειαζόμαστε 20.000 γιατί και το Μογκαντήσου πρέπει να το κρατήσουν αλλά και όλη τη χώρα και ιδίως ε, το Κισμάγιο, το λιμάνι αυτό στο Νότο. Και η Αφρικανική Ένωση συνέχεια μας λέει ότι χρειάζονται 20.000 άτομα. Άρα χρειάζεται και χρηματοδότηση. Εγώ δεν μπορώ να ε, έρθω σε αντίθεση, γιατί αυτοί νομίζω ότι ξέρουν καλύτερα τις ανάγκες τους για τη Λιβύη. Αυτό το contingency plan πράγματι το έχουμε υπόψη μας και το κρατάμε και αν χρειαστεί ποτέ θα μπορούσαμε ε, να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια των κρατών. Στη στιγμή προς το παρόν κρατάμε στο συρτάρι αυτό το σχέδιο. Το θέμα είναι να δούμε αν υπάρχει κατάπαυση του πυρός και αν υπάρχει κατάθεση των εξοπλισμών. Γιατί υπάρχει κίνδυνος και με κάποιους ε, πυράβλους, ε, εδάφους που μπορεί να εξαφανιστούν. Πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει, ίσως η στρατιωτική θα δούμε. Και τελευταίο ερώτημα. Ψήφισμα 1325, πολύ σημαντικό ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών. Ε, γιορτάσαμε τη δεκαετία του επέτειο για το ρόλο των γυναικών συγκεκριμένα και τη συμμετοχή τη συμμετοχή, τη σημαντική συμμετοχή των γυναικών στην πρόληψη και τη βελτίωση. Κάναμε την ανάλυση μας του τι έχουμε κάνει εμείς εδώ και 10 χρόνια και νομίζω ότι πολλά έχουν γίνει σε πολλούς τομείς. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή. Έχουμε 15 ειρηνευτικές αποστολές σήμερα. Τις τρεις τις διευθύνουν γυναίκες. Στην Κύπρο, στο Νότιο Σουδάν, τέσσερις. Λιβέρια, Λιβέρια και Τιμόρ. 4 στις 15 λοιπόν τις διευθύνουν γυναίκες. Πριν από 7 χρόνια μια Φιλανδή ήταν μόνο μία όμως αποστολή. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πρώτο παράδειγμα. Δεύτερο, θέλουμε να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αστυνομία. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Ίσως είναι πιο δύσκολο στο στρατό, των διαφόρων χωρών. Είναι γύρω στο 3% συμμετοχή κατά μέσο αλλά στην αστυνομία θέλουμε να φτάσουμε στο 20% συμμετοχή γυναικών μέχρι το 2014. Στην αστυνομία, επαναλαμβάνω. Οι Ευρωπαϊκέ χώρε, οι Ευρωπαίοι, φυσικά είναι καλοδεχούμενοι, ευπρόσδεκτοι. Και όπως και η κυρία Γκόμες, έχουμε μια αστυνομική, ε, ειδική ε, γυναικεία ομάδα στη Λιβυρία που δίνει το καλό παράδειγμα και στο από τον Μπαγκλαντές γυναίκες μόνο στην ΑΕΤ, παραδείγματα πολύ θετικά. Γιατί δίνουν το παράδειγμα και στις ε, χώρες αυτές, στη Λιβυρία, που το είδε και η Λιβυρία έχει αυξήσει τον αριθμό των ε, ε, αστυνομικίνων. Και στις προς προσφύγων στον Ταρφούρ και αλλού οι γυναίκες έχουν μια πολύ πιο άμεση πρόσβαση με τα παιδιά και τις γυναίκες εκεί και γενικώ με τα θύματα κακοποίησης. Οπότε προσπαθούμε να αυξήσουμε τον αριθμό τους. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Και ένα τελευταίο σχόλιο, ένα τομέα στον οποίο βλέπουμε ότι δεν είχαμε σημειώσει μετά την ψήφιση του 1325 μεγάλη πρόοδο, συμμετοχή γυναικών στη διαμεσολάβηση ε, σε περίπτωση συγκρούσεων. 6 με 7% ε, είναι οι γυναίκες διαμεσολαβήτριες είναι ένα τομέα που προσπαθούμε εμείς όσο μπορούμε στον Darfur, είμαστε διαπραγματεύσει μεταξύ επαναστατών και κυβερνητικών δυνάμεων και προσφύγων και προσπαθούμε να αυξήσουμε το διαμεσολαβητικό ρόλο των γυναικών, αλλά εκεί έχουμε πάρα πολύ ακόμη ε, πρόοδο να επιτελέσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λερουά. Σας ευχαριστούμε για όλες αυτές τις ε, πληροφορίες και για τα σαφή μηνύματα τα οποία απευθύνατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα εξοπλισμού και προσωπικού που χρειάζεστε. Επίσης, πολύ θεωρητικά αντιμετωπίζουμε το θέμα των battle group. Ε, είναι πάρα πολύ καλό να ακούμε προτάσεις για συγκεκριμένη χρήση των battle group. Έχουμε δύο λεπτά. Ο συνάδελφος θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Λέει ο κύριος Γιάννης. Θέλω να ρωτήσω και δεν πρόκειται εδώ για αρρωστημένη περιέργεια. Εμένα με, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παρουσίαση του κυρίου Λερουά. Αλλά στην ημερήσια διάταξη τον κύριο Λερουά εδώ τον εμφανίζουμε πρώην γενικό γραμματέα, πρώην διευθυντή κτλ. Οπότε θέλω να ξέρω τι είναι σήμερα. Ήταν τόσο ενδιαφέροντα όλα όσα αυτά μας είπε που όλα τούτα τα πρώην πρώην Ε, λοιπόν, ήθελα να ξέρω τι είστε. Είστε υπάλληλο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, του ΟΗΕ, σίγουρα είστε ένα Γάλλο υπάλληλο, αλλά ποιο είναι ο ρόλο σα σήμερα, γιατί θα θέλαμε να σα ξανακούσουμε στην Επιτροπή μα. Καλή ερώτηση. Εγώ είμαι Γάλλος υπάλληλος, αποσπασμένος στον ΟΗΕ για οικογενειακούς λόγους δεν ανανέωσα αυτή τη διετή θητεία για, ε, τέσσερα, ε, για τέταρτη φορά. Εγώ είμαι σύμβουλος του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα έχω άλλου είδους διεθνείς αρμοδιότητες. Εγώ πάντως σήμερα είμαι σύμβουλος του Ελεγκτικού συνεδριού στη Γαλλία, το στρες εκεί είναι λιγότερο ισχυρό. Για τα battle group όμως να σας πω, στη συζήτηση που είχε γίνει, που έγινε, η εντύπωση ήταν ότι τα battle group στοιχίζουν ακριβά. Αλλά πολλές χώρες ήδη έχουν ε, συγκροτήσει τα battle ε, group τους. Οπότε το να τα καταστήσουν επιχειρησιακά πλέον στοιχίζει πολύ λιγότερο. Τα battle group ε, τα συζητήσαμε προηγουμένως σχετικά με τις οικονομίες που θα μπορούσαμε να είχαμε στην Ευρώπη από την αναδιοργάνωση των στρατευμάτων μας. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ τον κύριο Σαλμή να έρθει. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας. Έχω την ευχαρίστηση να υποδέχομαι σήμερα τον κύριο Σαλμή, ο οποίος από τον Φεβρουάριο είναι διεύθυντης του ΣΥΤΧΕΝ, αποσπασμένος παρά την υπάτη εκπροσώπου. το ΣΥΤΣΕΝ θεωρείται ε, έχει μάλλον μια παραμορφωμένη εικόνα στους ε, βουλευτές θεωρείται ως η, η ευρωπαϊκή ΚΥΠ. Θα θέλαμε να μας το εξηγήσετε καλύτερα. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η θέση σας σε αυτό το νέο οργανόγραμμα εξωτερικής δράσης, ε, τι επικάλυψη μπορεί να υπάρχει με άλλους οργανισμούς που εργάζονται στον τομέα της intelligence, με την Ευρωπόλ και άλλους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Συναντήσατε ήδη τους βουλευτές στην ΛΥΜΠΕ, αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στην Επιτροπή ΣΕΝΤΕ. Έχετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη του να σας ευχαριστήσω καταρχάς για την ευκαιρία που μου δίνετε να απευθυνθώ στην υποεπιτροπή σας για θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα και μάλιστα πολύ παραγωγικά, ώστε να διαφωτίσουμε λίγο για το τι γίνεται ακριβώς ε, στην ε, κατάσταση στην Ευρώπη και τι έμαθα εγώ τους τελευταίους 8 μήνες που, είμαι, που βρίσκομαι εκεί, γιατί υπάρχουν πολλές φήμες, πολλές παρανοήσεις για το τι κάνουμε γενικώ. Όπως είπε ο Πρόεδρος, δεν είμαστε μυστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά έχουμε στρατηγικό ρόλο στο να παρέχουμε ε, υποστήριξη σε μυστικές υπηρεσίες και σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε θα προσπαθήσω να σας διαφωτίσω για το τι ακριβώς κάνουμε. Θα ξεκινήσω πολύ σύντομα για την αποστολή του Σίτσεν. Θα σας πω λίγα πράγματα για, το, για την ιστορία του και για το τι κάνουμε σήμερα και τι ακριβώς, με τι ακριβώς ασχολούμαστε. Από αυτό θα ξεκινήσω και βεβαίως ευχαρίστω θα σας απαντήσω εάν έχετε ερωτήσεις. Η αποστολή μας. Για να διατηρήσουμε μια ασφαλή Ευρώπη σε έναν καλύτερο ε, τρόπο, όπως αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ε, σωστές πληροφορίες έτσι ώστε να λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Όπως γίνεται παντού στον κόσμο, σε κάθε κράτος είναι μια γενική αλήθεια αυτή. Το Citizen από το 2002 παρέχει τέτοιες πληροφορίες και αναλύσεις. Η αποστολή του είναι να δώσει την ανάλυση των, ε, πληροφοριών, να ενεργοποιήσει την ε, ε, ετοιμότητα μέσω της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων και της υπάτου προσώπου καθιάστων. Το Citizen επίσης επικεντρώνεται σε ευαίσθητες γεωγραφικές περιοχές, σε, στην στην διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και σε άλλες παγκόσμιες απειλές το ΣΥΤΣΕΝ προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε, διάφορες, ε, σε διάφορα ε, σε διάφορες υπηρεσίες και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και ε, μεμονωμένα στα κράτη-μέλη. Η δημιουργία του ΣΥΤΣΕΝ συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Ασφαλείας και τη δημιουργία της θέσεως ε, του ΙΠΑ του Αρκοπροσώπου το 1999. Οι δυνατότητες αντιμετώπισης κρίσεων και η ανάπτυξη και πολιτικών και, και στρατιωτικών επιχειρήσεων αποστολών έδειξε ότι η γενικότερη δομή, χρειαζόταν μια διαφορετική δομή για την ανάλυση των πληροφοριών. Η, τα γεγονότα τη 11 Σεπτεμβρίου και η, ε, απειλή, παγκόσμια απειλή τη Τρομοκρατία τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει όντω καλύτερη ανάλυση των ε, μυστικών πληροφοριών ώστε να υποστηριχθεί η Ευρώπη. Γι' αυτό το 2002 δημιουργήθηκε το Citizen ω ε, διεύθυνση τη γραμματεία του Συμβουλίου άμεσα συνδεδεμένη με, την υπηρεσία τη ΥΠΑ εκπροσώπου. με προσώπου από τα κράτη-μέλη οι οποίοι είναι ε, αποσπασμένοι στο Σίτσεν. Το 2005 το Σίτσεν ενισχύθηκε από την άφηξη μιας ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων από τις ομάδες αντιτρομοκρατίας που σημαίνει από τις ε, υπηρεσίες ασφάλειας ε, των κρατών μελών και την Ελβετία και την Ορβηγία. Αυτό ε, μας βοήθησε να παράσχουμε στην EAS και στο Συμβούλιο αξιολόγηση των απειλών με βάση τις πληροφορίες που είχαμε από τις εθνικές υπηρεσίες. Από το 2007 το ΣΥΤΣΕΝ εργάζεται μαζί με, την, ε, με, το, στρατιωτικό, με το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια, ε, σε μια ε, μονάδα την SIAC. Όλες οι αξιολογήσεις που εκδίδονται στα κράτη-μέλη είναι παράγωγα κοινών προσπαθειών στα πλαίσια της ΣΥΑΚ μετά την ε, θέση ισχύ τη ε, Συνθήκη Λισαβόνα, το 1ο Δεκέμβριο του 2009, η Σίτσεν ε, ετέθη στην αποκλειστική ευθύνη τη υπάτου προσώπου τη Κάθη Άρστον. Λίγα λόγια τώρα για τις βασικές λειτουργίες και τα καθήκοντα του Σίτσεν. Η βασική λειτουργία είναι να παρέχει αποκλειστικές πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες αλλού στην είπατε εκπρόσωπο ή στην αντιπρόεδρο και στο, στην, πολιτική, στην Επιτροπή Πολιτική και Στρατιωτική με βάση τις ε, συμβολές των κρατών μελών ε, και των υπηρεσιών ασφαλείας τους. Δεύτερον, να παρέχει αξιολόγηση και ενημέρωση, καθώς επίσης και μια, ένα φάσμα προϊόντων που βασίζονται στην ε, ασφάλεια και μέσω open source, στην ΥΠΑΤΗ, και στην EAS, για, διάφορες, ε, για, τις, ε, για την λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά τα, την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και, καθώς, και των κρατών μελών. Τρίτον, να δρά ως σημείο, μοναδικό σημείο εισόδου των πληροφοριών μέσω των ε, υπηρεσιών ασφαλείας των κρατών μελών. Και τέταρτον, να βοηθάει τον ε, πρόεδρο του, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον πρόεδρο της Επιτροπής στην εξάσκηση των ε, καθηκόντων τους στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων. Τέλος, παρόλο που έτσι όπως έχει η κατάσταση τώρα το Citizen ε, αποτελεί έτσι ένα ε, πρόγραμμα που εξακολουθεί να εκτιλίζεται. Αυτά που σας παρουσιάσαμε ήδη χτες ε, αναφέρουν την δομή του κτλ. Αλλά θα πρέπει να πω ότι αυτό είναι μια δουλειά που εξελίσσεται και το τελικό αποτέλεσμα της θα ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες ή ίσως και τον επόμενο μήνα, έτσι ώστε να γνωρίζουμε. Αλλά οι βασικές λειτουργίες του Citizen είναι η ανάλυση των πληροφοριών και από την δημιουργία του. Το Citizen αυτό κάνει, δίνει στρατηγικές α, αναλύσεις για την διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα πράγμα που πρέπει να πω οπωσδήποτε είναι ότι το Citizen δεν είναι επιχειρησιακό κέντρο ή υπηρεσία ασφάλειας ή μυστικών υπηρεσιών. Λέγοντας αυτό, θέλω να πω ότι δεν έχουμε δυνατότητες τέτοιε συλλογή πληροφοριών όπως τα κράτη-μέλη και οι δικές τους υπηρεσίες πληροφοριών. Δεν εμπλεκόμεθα με κανένα τρόπο σε κανένα είδους ε, επιχειρήσεις ούτε στην Ευρώπη ούτε στις τρίτες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι κάτι σημαντικό και μας διαχωρίζει σαφώς από τις επιχειρήσεις που γίνονται από τα κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες τους και σύμφωνα με την νομοθεσία τους. Δεύτερον, δεν έχουμε το δικαίωμα συλλογής προσωπικών δεδομένων, που σημαίνει ότι πρέπει οι αξιολογήσεις μας να γίνονται σε ένα πολύ στρατηγικό επίπεδο, που κατά την άποψή μου είναι ακριβώς ο ρόλος που θα πρέπει να επιτελεί το Citizen και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να, ε, εφαρμόζουμε τα, όσα, τα καθήκοντά μας. Τέλος, οι υπηρεσίες μας και οι πηγές που χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι πρέπει. Για τα προϊόντα. Η ραχογκαλιά των ε, δραστηριοτήτων Citizen, ε, ας πούμε, αξιολόγηση καταστάσεων, situation assessment, βασίζονται σε, μια, σε έναν κατάλογο ε, ο οποίο ενημερώνεται κάθε 6 μήνε, στρατηγικά έγγραφα τα οποία βασίζονται επίση σε βασικέ πληροφορίε από τι πληροφορίε που λαμβάνουμε από τι υπηρεσίε πληροφοριών των κρατών μελών, εκπονούνται. Κάνουμε αξιολογήσει κινδύνων με βάση του κινδύνου ε, και με τη βοήθεια των ε, σχετικών εμπειρογνωμόνων από την ε, εκάστοτε χώρα. Κάνουμε κάποιου ελέγχου, πρώτε αντιδράσει μετά από κάποιο συμβάν, μπορεί να είναι μια τρομοκρατική επίθεση, όπω α πούμε στο Όσλο τον Ιούλιο, ή μπορεί να είναι κάτι σαν τα πιο πρόσφατα γεγονότα που γίνονται στην ε, Βόρεια Αφρική. Κάνουμε ειδικές, ε, ειδικέ εκθέσει για την παρακολούθηση μιας κατάστασης ή ένα θεματικό έγγραφο που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα θέματα επίκαιρου ενδιαφέροντο, Ας πούμε, μια ε, έκθεση για, την ακροδεξιό, για τον ακροδεξιό εξτρεμισμό στην Ευρώπη μετά το συμβάν στο Όσλο. Επίσης κάνουμε ενημερώσεις εβδομαδιαίες όπου επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την εβδομάδα με κάποια μικρή ανάλυση των ε, πληροφοριών, των μυστικών πληροφοριών. Πέρα από αυτό έχουμε πολλά ε, εργαλεία ε, online ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την δουλειά της υπάτου προσώπου και άλλων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να πω ότι επίσης ε, έχουμε πάρα πολύ καλές ε, σχέσεις με το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιοι από τους συναδέλφους μου έχουν ενημερώσει τις αντιπροσωπείες των, του Κοινοβουλίου που πηγαίνουν σε κάποιες περιοχές όπου υπάρχουν κρίσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να παρέχουμε και σε εσά τις απαραίτητες πληροφορίες για να μπορέσετε να έχετε μια εις βάθος αξιολόγηση της κατάστασης στην χώρα στην οποία πρόκειται να, την οποία πρόκειται να επισκεφτείτε. Και χαίρομαι που αυτό έτυχε θετικής αντιμετώπισης και από τον. Κοινοβούλιο και χαίρομαι που μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την αγαστή συνεργασία. Λίγα λόγια τώρα για τα προϊόντα και τις πηγές. Όπως είπα, η βασική πηγή είναι η, κοινωνία μυστικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δίνει αξιολογημένες πληροφορίες, τις οποίες χρησιμοποιούμε μετά εμείς στις δικές μας αξιολογήσεις. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε ευρέως διαθέσιμες ε, ε, πηγές όπως blog, ε, ιστοσελίδες, open source ιστοσελίδες κτλ. Επίσης, διπλωματικές εκθέσεις που έρχονται από τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αξιολογούμε και τις συγκρίνουμε με τις δικές μας πληροφορίες που έχουμε λάβει και από άλλες πηγές. Και όπως είπε ο Πρόεδρος στα αρχικά του σχόλια, συνεργαζόμαστε με το, κέντρο, το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λαμβάνουμε και από αυτούς πληροφορίες ό,τι αφορά την, ε, τις δορυφορικές εικόνες, ε, έχοντας υπόψη βεβαίως ότι δεν παρέχουμε και ούτε θα παρέχουμε στο μέλλον τακτική ή ε, ε στρατιωτική ενημέρωση από τη δική μας την πλευρά. Απλώς χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία. Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ευχαρίστω να απαντήσω ή να ακούσω και σχόλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ που διευκρινίσατε τον τρόπο λειτουργίας του ε, κέντρου. Όπως ε, το είπα και εγώ πριν ε, στην παρουσίασή μου υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση για το πώς το κέντρο λειτουργεί και πού τοποθετείται ακριβώς. Ε, έχω μία ερώτηση σχετικά με τη λειτουργία. Αναφέρατε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν διαθέτεται ίδιους πόρους. Δεν διαχειρίζεστε ίδιους πόρους, εξαρτάστε από αυτό που σας χορηγούν οι υπηρεσίες των κρατών μελών. Γνωρίζουμε καλά ότι ορισμένες υπηρεσίες ασφάλειας των κρατών μελών μπορούν να βρίσκονται σε ανταγωνιστική θέση μεταξύ τους για την αξιολόγηση κρίσεων, προσώπων κλπ. Ποια, πώς γίνεται η διαιτησία μέσα στο κέντρο διαχείρισης των Ας πούμε έχουμε την Ευρωπαϊκή Αποστολή στα Βαλκάνια. Πώς γίνεται η αξιολόγηση ε, τις, ε, πώς οι εκθέσεις των διαφόρων μυστικών υπηρεσιών, αγγλική, γαλλική κλπ. μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους. Στο Σίτσεν ποιος έχει την τελευταία λέξη, υπάρχει ένας χώρος έκφρασης των διαφωνιών για να μπορείτε να έχετε μία πληρέστερη εικόνα των πληροφοριών. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο προς τα έξω εσείς εξετάζετε και τις πληροφορίες που σας έρχονται από τις εξωτερικές αντιπροσωπείες. Οπότε φαίνεται τελικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται πολύ πιο σημαντικές πληροφορίες από ότι οι μυστικές υπηρεσίες των κρατών μεμονωμένα. Ε, αυτό ξεπερνάει τα όρια των αρμοδιοτήτων των κρατών μελών. Επειδή ακριβώ έχετε αυτές τις περισσότερες ε, μυστι... Ε, απόρριτες πληροφορίες στη διάθεσή σας, αυτό δεν σας δημιουργεί τον πειρασμό να αυτονομηθείτε ως προς τη διαχείριση της πληροφορίας. Ο κύριος Πάσκου ήθελε το λόγο. Ε, ανταγωνισμός με τον κύριο Πάσχου. Καταλαβαίνω ότι δεν είστε μια υπηρεσία πληροφοριών, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είστε. Αλλά θέλω να ρωτήσω πώς λειτουργεί η μονάδα σας, διότι όλοι. πρημοδοτούμε την ανάλυση. Ρωτώ λοιπόν εσείς πώς ε, τα αναλύετε τα έγγραφά σας, ε, με ποια οπτική, τη δική σας ή των κρατών μελών. Πώς συνεργάζεστε με τις εσωτερικές υπηρεσίες, ε, ζητείτε ε, δικές σας πληροφορίες ή τομεακές πληροφορίες, διότι σήμερα είναι της μόδας να ζητάει κανείς ε, αναλύσεις ε, ιδιωτική intelligence. Συνεργάζεστε με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για αυτά τα ζητήματα. Πώς προσλαμβάνετε εσείς τους εμπειρογνώμονες στην ε, μονάδα σας. Και τελευταίο, επειδή είστε στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, τι έχετε κατά νου για να βοηθήσετε τις αποστολές. σχεδιάζετε να έχετε μία υποστήριξη για τις αποστολές. Ε, ευχαριστώ. Κύριος Πάσχου. Ευχαριστώ. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επέτρεψα στην κυρία να προηγηθεί δεν είναι μόνο επειδή είμαι εξορισμού ευγενής, αλλά και γιατί ήξερα ότι θα θέτατε ερωτήματα που θα έθετα και εγώ και άρα έπρεπε να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ μας. Τέλος πάντων, εσείς εδώ ουσιαστικά έχετε το πλεονέκτημα, ας πούμε, σε σχέση με τα εθνικά κράτη, ότι μπορείτε τις πληροφορίες, το intelligence, αλλά και τις εκτιμήσεις που έχετε από πολλές πηγές να τις συγκεντρώνετε. Έχετε feedback που μπορείτε να κάνετε προς τις άλλες χώρες Δηλαδή, όλοι συνεισφέρουν σε εσά, κάνετε εσεί μια σύνθεση, μια ανάλυση την οποία μετά την ανατροφοδοτείτε σε όλε τι χώρε. Γιατί ξέρετε, μπορούν και αυτέ να συζητήσουν μεταξύ του, μεν, αλλά το πλεονέκτημα που έχετε εσεί είναι ότι ουσιαστικά ενσωματώνετε, ενώνετε πολλέ πηγέ. Όταν τώρα έχουμε να κάνουμε με αυτό το είδος αξιολόγησης που έχετε, πού βασίζεται στη δική σας ικανότητα εκτίμησης και ανάλυσης. Ή ζητείτε όχι μόνο πληροφορίες αλλά και εκτιμήσεις από τα κράτη. Πώς λειτουργεί ακριβώς. Ευχαριστώ. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σύντομα ερωτήματα. Τα δύο πρώτα βέβαια ετέθησαν ήδη από τον πρόεδρο Ντανζό. Για την ε, τρομοκρατία. Στα διάφορα φόρουμ και μελέτες ακούγεται συχνά ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εξής λύση ότι θα έπρεπε να πνίξουμε τον, την τρομοκρατία στα γενοφάσκια της. Πρέπει πάντοτε να έχουμε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση του Μαλή για να, να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία στην περιοχή του Σαχέλ. Το ΣΥΤΣΕΝ συμμετέχει σε αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε λύσεις στα προβλήματα τρομοκρατίας επιτόπου. Και όσον αφορά στη στρατιωτική συνεργασία, έχουμε μια άλλη πρόταση που έγινε, πολλές, διατυπώθηκε πολλές φορές, Όταν υπάρχει κρίση θα ήταν καλό να συνεργάζεστε με τους στρατιωτικούς ε, φορείς ε, των χωρών της Ένωσης. Εσείς λαμβάνετε τώρα πληροφορίες από τα κράτη-μέλη, κάνετε συνθέσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. Έχετε όμως ένα περιθώριο χειρισμών όταν αυτές οι πληροφορίες είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Ή παράλληλες ή ελλειπείς όταν έχετε πληροφορίες που αφορούν σε τρίτες χώρες και εσείς έχετε την απαγόρευση της τρίτης χώρας να διαβιβάσετε αυτές τις πληροφορίες. Τι κάνει το Citizen στην προκειμένη περίπτωση, τηλεφωνεί στο κράτος μέλος και ζητάει παραπάνω πληροφορίες. Άλλη ερώτηση. Θα έχετε μία επιχειρησιακή εντολή για το μέλλον. Διότι τίθεται το ερώτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει την υπηρεσία, τη δική της υπηρεσία πληροφοριών. Ας πούμε η Ευρωπόλ πολλές φορές μας λέει ότι θα χρειαζόταν να έχει επιχειρησιακή εντολή διότι αυτή η έλλειψη εντολής αποτελεί ένα κενό και ένα εμπόδιο για τις δραστηριότητες Ευρωπόλ. Φαντάζομαι ότι το αντίστοιχο θα είναι πρόβλημα και για το Σίτχεν. Εσείς παίρνετε όλες τις πληροφορίες, κάνετε και μία ανάλυση τάσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να μας μιλήσετε για την ριζοσπαστικοποίηση για παράδειγμα των μουσουλμάνων ε, και τι γίνεται με την ρίζο ε, σπαστικοποίηση της τρομοκρατίας και την διάσπασή της μετά το θάνατο του Μπιν Λάντεν. Στις διάφορες περιοχές του κόσμου παρακολουθείτε εσείς όλες αυτές τις τάσεις και δεν μιλάω εδώ μόνο για, δεν μιλάω μόνο για την Αλκαΐδα, μιλάω για τις ε, νέες αυτόνομες ομάδες. Επίσης, ε, τι γίνεται με την άκρα δεξιά και την άκρα αριστερά. Τις ίδιες ερωτήσεις είχα, ρωτήσει, κάνει και στην Ευρωπόλ. και η Ευρωπόλ είπε ότι η ακραία οι ακραίοι ριζοσπάστες ε, επηρεάζουν τους πάντες. Ε, χθες ε, στην Λίμπε συναντήσαμε ένα ίδρυμα από τη Γενέβη, την ΛΙΚΑΠ, που έχει, έχει φτιάξει μία μελέτη στην οποία συμπεριλάβωνε η Ευρωπόλ, η ΣΥΤΧΕΝ, και θέλει να μας προτείνουν να φτιάξουμε μία κοινοβουλευτική επιτροπή, θέλουν ένα screening. Υπάρχει βέβαια μία αντίφαση σε αυτή τη μελέτη. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σαλμί έχει μάθει σχετικά με αυτή τη μελέτη. Λοιπόν, ε, τι λέτε εσείς, ε, είναι η υποεπιτροπή της ε, ΛΥΜΠΕ που ασχολείται με το θέμα. Φαντάζεστε ότι ίσως η ΣΕΝΤΕ δεν είναι πιο αρμόδια. Οι ερωτήσεις ε, προς τον κύριο Σαλμή αφορούν στην οργάνωση και την μεθοδολογία και για τα θέματα τρομοκρατίας, αντιμετώπιση και αντιμετώπιση της ε, είναι εκτός θέματος. Ο κύριος Χερνάουζερ. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Ένα ερώτημα έχω για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η κοινοβουλευτική έλεγχη ακόμα είναι στα σπάργανα. Η συζήτηση ξεκινάει, έχουμε μία κρόαση για το θέμα αυτό. Χτες έγινε, παρουσιάστηκε μία ε, μελέτη στην Επιτροπή Λίμπε και μία σύσταση είναι να υπάρξει ανα, μεταρρύθμιση όλων αυτών των θεμάτων. Η σύσταση λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει θεσμική συμφωνία με την EAD για μια γενική πρόσβαση σε υποθέσεις όπου και ο ελεκτής από μόνος του μπορεί να αποφασίσει τι είναι χρήσιμο από τα στοιχεία για τον έλεγχο και τι όχι θα με ενδιαφέρε να μου πείτε τη γνώμη σας. Τι, γνώμη έχετε για την ε, γενική αυτή πρόσβαση σε τέτοιες ε, υποθέσεις ε, και τι άποψη έχετε για την συμφωνία αυτή μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργάνων και του EAD. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στάτσιν. Thank you, Ευχαριστώ. Έχω και εγώ κάποια σύντομα ερωτήματα. γιατί κάποια στοιχεία δεν τα βλέπω στο κείμενο. Μιλήσατε για οργάνωση και είπατε ότι μπορείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείτε να είσαστε ε, πολύ αποτελεσματικοί παρά τον, τον πολύ αυστηρό προπολογισμό σας. Ε, πόσα, τι ποσοστό στελεχών έχετε, τι ακριβώς αριθμό υπαλλήλων έχετε, ποιος είναι ο προπολογισμό σας, σας ικανοποιεί, ε, βλέπετε να υπάρχουν ε, ανάγκες για διεύρυνση, ε, είναι για αύξηση της ποιότητας και ένα ακόμη ερώτημα. Συλλέγετε εσείς τις πληροφορίες από τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είναι σε θέση να θέσουν σε εσά ερώτημα, να ζητήσουν από εσά πληροφορίες. Ευχαριστώ. Merci, Madame Κυρία Γκόμες. Uh, Ευχαριστώ. Να ρωτήσω κι εγώ. Σημείωσα αυτό που είπατε, ότι δεν ε, συμμετέχετε σε κανένα είδου επιχειρήσει. Μπορείτε όμω να στείλετε το προσωπικό σας επιτόπου, α πούμε, να, για μια έτσι καταγραφή των αναγκών για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο, αν γινόταν κάτι τέτοιο. Επίση άλλο ένα ερώτημα, νομίζω τέθηκε ήδη. Μπορείτε εσείς να πάρετε την πρωτοβουλία και να επικεντρωθείτε σε μια, σε μια περιοχή, σε μια απειλή και να την προωθήσετε αυτή την ιδέα σας ως, ε, στην ύπατη εκπρόσωπο ή περιμένετε από την ύπατη εκπρόσωπο να σας, ε, να σας αναφέρει τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε. Επίσης αυτό το, αυτός ο κατάλογος που έχουμε εδώ λέει ότι παρέχετε υπηρεσίες σε διάφορες ε, υπηρεσίες, ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφέρονται διάφορα η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, η κοινή πολιτική, εξωτερική πολιτική. Στην παρούσα φάση ε, στις ε, εντάσεις που υπάρχουν μεταξύ Κύπρου και ε, Τουρκίας. Ποιες ακριβώς είναι οι συνέπειες. Έχουν, επίσης έχουν εξαφανιστεί 10.000 τμήματα πυράβλων στη Λιβύη. Τι γίνεται. Επίσης, οι Κινέζοι έχουν ξεκινήσει ένα, μια επιχείρηση αγορών στην Ευρώπη, τεχνολογίας μπορείτε εσείς να παρέμβετε σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, ε, έχετε επαφή με τις ε, μυστικές των κρατών μελών και προφανώς βασίζεστε και σε αυτές εν μέρη. Η δική σας κρίση της απόδοσής τους ποια είναι. Και δεν εννοώ την αντιπαλότητα που μπορεί να υπάρχει, αλλά πραγματικά την απόδοσή τους. Ε, στην χώρα τους. Εσείς μπορείτε να την κρίνετε, γιατί προφανώς και εκεί υπάρχουν ε, και εσωτερικά υπάρχουν ανταγωνισμοί. Και κάποιες ίσως αποτυχίες ή κάποια προβλήματα. Μπορείτε να κρίνετε εσείς αυτό το, αυτή την κατάσταση ίσως να ήταν ε, και χρήσιμο για την αντιμετώπιση ας πούμε, της θερμοκρατίας λοιπά Ευχαριστώ κύριο Λαντσμπέργκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα κάποιες περισσότερες διευκρινήσεις σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του κέντρου του ΣΥΤΣΕΝ για τις επιχειρήσεις, τις αποστολές. Η αποστολή του είναι να παρέχει αναλύσεις πληροφοριών και τα λοιπά σε ένα άτομο λέει και σε ένα γραφείο. Mission, αποστολή, αυτό λέει. Και μετά, πέραν της αποστολής, διατίθενται και υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες, ακόμη και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται ως πελάτες, τη βλέπω εδώ. Λέει όμως ότι μπορεί να παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες υπό μορφή ε, εκτιμήσεων ρουτίνας κάθε 6 μήνες και υπό τη μορφή ενημερώσεων, briefings, κατόπιν ειδικού αιτήματο, ενδεχομένως. Αλλά όχι αποκλειστικές πληροφορίες, γιατί οι αποκλειστικές πληροφορίες είναι μόνο για ένα άτομο, ένα γραφείο. Μετά, λέει, ταξινομημένες, διαθεσμένες πληροφορίες οι... Ε, άλλα στοιχεία έρχονται από τα κράτη-μέλη προς το όχι όμως προς τα κράτη-μέλη. Επομένως, το ερώτημά μου το εξής. τα κράτη-μέλη και οι κυβερνήσεις με ποιο τρόπο ή με ποια μορφή θα μπορούσαν να λαμβάνουν πιο ευαίσθητες ή πολύτιμες πληροφορίες για κάτι το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ε, κίνδυνος για αυτά, τα κράτη-μέλη δηλαδή. Λέτε παροχή αναλύσεων πληροφοριών, παρακολούθηση, αξιολόγηση. σε λεπτούς ευαίσθητους τομείς και για τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Λέτε. Πώς να εννοήσουμε αυτή τη διάδοση οπλομασικής καταστροφής. Παραδείγματος χάρη, σε ό,τι αφορά το Καλίνιγκραντ, την περιοχή του Καλίνιγκραντ, εκεί τι έχουμε, διάδοση ή όχι. Υπάρχουν εκεί όπλα μαζικής καταστροφής. Και είναι, ξέρετε, πολύ κοντά η περιοχή αυτή στην Πολωνία και στη Σουηδία και Και κάτι άλλο. Πύραυλοι, βλήματα που μπορούν να πλήξουν πυρηνικά εργοστάσια, αν χρειαστεί. Υπερήφανα το ανακοίνωσε ο ύπατος διοικητής του Ρωσικού στόλου στο Καλίνιγκραντ. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε βόμβες, έχουμε πυράβλους που μπορούν να στοχεύσουν και να πλήξουν πυρηνικούς σταθμούς. Υπάρχουν δηλαδή βόμβες εκεί και μπορούμε και εμείς να εξάγουμε, αν θέλετε, αυτές τι βόμβε. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα, η Ρωσία φτιάχνει δύο βόμβες ενδεχόμενες τέτοιες στα σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούνται αυτοί οι πύραυλοι όπλα μαζικής καταστροφής. Αν στραφούν κατά πυρηνικών σταθμών. Σε συνδυασμό με αυτό. Και ποιο είναι το όραμα, θέλετε, ποια είναι η σκέψη ε, του κέντρου επιχείρησης του Σίτσεν σε σχέση με κάτι τέτοιο και αν έχετε πληροφορίες. Θα μπορούσατε να ενημερώσετε εσείς τα κράτη-μέλη. η κυρία Άστον. Euh, Νομίζω έχετε πολλά ερωτήματα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι έλαβα πολλά ερωτήματα και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα. Να ξεκινήσω εδώ με την αντιπρόεδρο, η οποία πρέπει να φύγει όμως. Λοιπόν, ή μάλλον πρώτα να μιλήσω λίγο για τη διαδικασία Δηλαδή, αν με δική μας πρωτοβουλία κάνουμε κάτι ή αν έχουμε έτοιμα από κάποιο πελάτη, τέλος πάντων, πώς λειτουργούμε. Να σας πω ότι πρώτα απ' όλα ε, είναι συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή, μπορούμε να αναλάβουμε ίδια πρωτοβουλία, να δούμε κάποια από τα θερμά σημεία, από τα hot spots, τα οποία θα πρέπει για το οποία μάλλον θα πρέπει να δώσουμε πληροφορίες στους πελάτες μας. Ιδίω όμως σε μακροχρόνιες ή μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις, Έχουμε αυτό το watch list. Κάθε έξι μήνες δηλαδή έχουμε αυτό το εγχείρημα, αυτή την άσκηση όπου εξετάζουμε κάποια θεματικά ζητήματα και περιοχές που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ να έχουν ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη ροή πληροφοριών, θα ήθελα να τονίσω ότι παρέχουμε τις εκτιμήσεις μας στις υπηρεσίες των κρατών μελών γενικά στα κράτη-μέλη. Δηλαδή λαμβάνουν ε, τα κράτη-μέλη οτιδήποτε εμεί κάνουμε. Είναι αμφίδρομη επικοινωνία. Και εγώ προέρχομαι από την υπηρεσία ενό κράτου μέλους και τα γνωρίζω. Πρέπει να υπάρχουν ανταλλάγματα. Φυσικά και δεν είναι υποχρεωτικό καμία υπηρεσία να μα δώσει το οτιδήποτε. Ουσιαστικά ε, η σχέση μα βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και θέλουμε να έχουμε και προστιθέμενη αξία και για τι υπηρεσίε των κράτων μελών και εν γέν για τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και παρέχουμε στα κράτη-μέλη τις δικές μας αναλύσεις και εκτιμήσεις. Για την πρόσληψη μου ένα ερώτημα, τις προσλήψεις. Οι περισσότεροι αναλυτές μας προέρχονται από τις υπηρεσίε των κρατών μελών. Έχουν μετατεθεί από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή έχουν προϋπηρεσία στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας τους και έρχονται σε εμά με απόσπαση για 2-6 χρόνια. Πέραν αυτού, Έχουμε και Ευρωπαίους αξιωματούχους οι οποίοι κάνουν και αυτοί αναλυτικό έργο και έχουμε βρει τρόπους με μπορούμε να έχουμε ανταλλαγή όλων των πληροφοριών. Όλοι όσοι εργάζονται στη, στο ΣΥΤΣΕΝ έχουν λίγο πολύ την ίδια πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που έρχονται από τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η βασική διαδικασία προσλήψεων, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά ε, τις θέσεις ADAST δημοσιεύονται οι προκηρύξεις με τον ίδιο τρόπο όπως οποιαδήποτε άλλη θέση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Φυσικά χρειάζεται έγκριση ασφαλείας ε, για οποιοδήποτε εργαστή στο SITCHEN, Security Clearance. Ποια είναι η διαδικασία. Όταν αρχίζουμε με μια εκτίμηση. Φυσικά έχουμε έτοιμα πληροφοριών από τα κράτη-μέλη και εξετάζουμε και τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας. Ποιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και θα μπορούσαμε να τις συλλέξουμε ε, από ανοιχτές πηγές. Και έπειτα ολοκληρώνουμε την αξιολόγηση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ενημερώνουμε βέβαια τους πελάτες, τους δίνουμε όλα τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ανοιχτέ πηγέ, πληροφορίε επίση και από τι υπηρεσίε, ερώτημα κυρίω του Προέδρου για τι διάφορε εκτιμήσει ε, των ε, υπηρεσιών των κρατών μελών. Νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κοινή ευρωπαϊκή αξιολόγηση όλων των διαφορετικών απόψεων των κρατών μελών. Αν συμβαίνει αυτό. Συχνά βέβαια δεν συμβαίνει, συχνά έχουμε συνεπείς ενεκτικές απόψεις που αλληλοευθυγραμμίζονται μεταξύ τους, αλλά ενίοτε συμβαίνει. Ο ρόλος του Σίτσεν είναι να προβεί σε μια αξιολόγηση ευρωπαϊκή, ενωσιακή θα έλεγα. Όχι δηλαδή να αναφέρει τη θέση ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους, αλλά να βασίζεται στα πραγματικά περιστατικά για οποιαδήποτε μεμονωμένη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες τώρα που λαμβάνουμε, και για να έχουμε λίγο μεγαλύτερη ανεξαρτησία από τις υπηρεσίε των κρατών μελών. Αυτό μας δίνει μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Να σας πω ότι εμείς ως Ιτσεν βέβαια εξαρτώμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίε των κρατών μελών. Είναι ένα αξιόπιστος εταίρος. Ταυτόχρονα βέβαια πρέπει να ενισχύσουμε και τις δικέ μα δυνατότητες όσο το δυνατόν περισσότερο. Και αυτό βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι σήμερα, όπως συχνά στο, χρόνο, χώρο των πληροφοριών, ο χρόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να δίνουμε πολύ γρήγορα πληροφορίες, ιδίω σε ό,τι αφορά τρέχοντα επίκαιρα ζητήματα και εκθέσεις. Εκεί πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν ευρύτερα δίκτυα πέραν των υπηρεσιών των κρατών μελών και πράγματι προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αποστολές για τους ειδικούς εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό επίσης είναι αμφίδρομο. Συνεργαζόμαστε και με άλλα θεσμικά όργανα, δηλαδή δεν περιοριζόμαστε στο πλαίσιο της ΕΙΕΔ, αλλά και με την Κομισιόν και με κάποιες γενικές διευθύνσεις της και κάποιους άλλους φορείς που είναι και αυτοί πολύ καλοί, πολύ σημαντικοί εταίροι για το Σίτσεν σήμερα. Ελπίζω η Κομισιόν να νιώθει το ίδιο. Ότι και εμείς δηλαδή μπορούμε να, να παράσχουμε προστιθέμενη αξία στην Κομισιόν. Για το feedback νομίζω απάντησα ήδη, δηλαδή ότι παρέχουμε και εμείς πληροφορίες. Και όχι μόνο στις υπηρεσίες των κρατών μελών, οι περισσότερε αξιολογήσει μα πηγαίνουν ε, και στην Πολιτική και Στρατιωτική Επιτροπή. Και οι πρέσβει δηλαδή ενημερώνονται, ενημερώνονται παίρνουν τι εκτιμήσει μα. Και κατά την προσωπική μου άποψη αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη έχουν, αν θέλετε, μια κοινή πλατφόρμα τουλάχιστον για να ξεκινήσουν τη συζήτηση επί ουδήποτε ζητήματος. Έχουμε εμείς ε, κάνει μια έκθεση έτσι θέλουμε να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία μας. Ετέθησαν κάποια ερωτήματα για την τρομοκρατία και τη στρατιωτική συνεργασία. Για τη στρατιωτική συνεργασία δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας, είναι οι συνάδελφοι από την ε, διεύθυνση που αφορά το στρατιωτικό προσωπικό και αυτοί ασχολούνται με τη στρατιωτική συνεργασία στα διάφορα μέρη του κόσμου. Βέβαια, εμεί σίγουρα του υποστηρίζουμε με τις δικές μας αναλύσεις πληροφοριών. Αλλά υπερβαίνει τις δικές μου γνώσεις το τι γίνεται σε αυτό το τομέα. Επίσης είπατε, σαφής εντολή του Σίτσεν, αλλά αναφέρθηκε και η Europol. Το Σίτσεν έχει σήμερα μια πολύ ξεκάθαρη εντολή. Θα πρέπει να σας πω. Και αν υπήρχε η επιθυμία ή η βούληση να προχωρήσουμε περισσότερο, ε, στο, να γίνουμε δηλαδή μια ευρωπαϊκή υπηρεσία πληροφοριών, ε, δεν είναι στη δική μου, στο δικό μου επίπεδο, δεν είναι το δικό μου κλιμάκιο που θα αποφάσισε κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχουν και πολιτικά και νομικά κολλήματα και εμπόδια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αν τεθεί κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω, όπως είπα, ότι είναι σαφής η εντολή μας. Στρατηγικές αναλύσεις κάνουμε για τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών, με βάση πληροφορίες που λαμβάνουμε από τα κράτη-μέλη. Πολύ σύντομα τώρα, για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την ουσία της δουλειάς μας, ε, όπως ε, μεταξύ άλλων το Καλίνιγκραντ. Να σας πω το εξής, ό,τι αφορά τη ριζοσπαστικοποίηση, ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Αυτό το εξετάζουμε εκ του σύνεγγυς και για του χρόνου προετοιμάζουμε και ένα πρόγραμμα για να έχουμε follow-up ε, του θέματος και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Οπότε θα έχουμε μια ευρωπαϊκή ανταλλαγή απόψεων για αυτά τα θέματα. Αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πρώτα απ' όλα, όπω σα είπα, έχω εργαστεί στα κράτη-μέλη στον τομέα των επιχειρήσεων και ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικά συστήματα σε ισχύ στα διάφορα κράτη-μέλη. Διάβασα, μάλιστα, την σύνοψη της μελέτης που ανέθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και θέλω να σας πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτα απ' όλα, δεν είμαστε επιχειρησιακός φορέας. Άρα διαφέρει λίγο ο δικός μας έλεγχος, η εποπτεία σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα. Αν πάντως χρειαστεί αυτό, εμείς είμαστε στα αρχικά στάδια, αλλά αν χρειαστεί, θα το αποφασίσουν οι φορείς λήψη αποφάσεων. Σε ποιο επίπεδο ε, θα μπούμε ως Σε Ό,τι αφορά τώρα τις εμπιστευτικές πληροφορίες, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι θα πρέπει να σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει οι πάροχοι των πληροφοριών και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες των κρατών μελών. Άρα περιορίζονται οι δυνατότητε που έχουμε για να διαδώσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Εάν υπάρχει συμφωνία με τα κράτη-μέλη ότι θα δοθεί η πληροφορία και δεν υπάρχει περιορισμός. Δεν θα ε, έχουμε καμιά πληροφορία, δεν θα έχουμε καμιά ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη, αν συμβεί κάτι τέτοιο. Οπομένως, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ξεκολουθούμε να είμαστε σε συζητήσεις με την ΕΕΔ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδίω ό,τι αφορά τι ειδικέ επιτροπέ, τα special committees. Και φυσικά και με πολύ πρόθυμο να παράσχω στι ειδικέ επιτροπές του Κοινοβουλίου στο δυνατόν περισσότερες πληροφορίε για να υπάρχει η βέλτιστη και η μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό είναι προ όφελο και του ΣΥΤΣΕΝ. Για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επειδή είμαστε τμήμα της ΕΙΕΔ, αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο έλεγχος που ασκείται στην ΕΙΕΔ έρχεται σε άμεση σχέση και με τι δραστηριότητε του Σίτσεν. Άρα υπάρχει από αυτήν την έννοια κοινοβουλευτικό έλεγχο σε κάποιο βαθμό. Μέγεθο και προπολογισμό. Είμαστε στην ίδια γραμμή του προπολογισμού με την ΕΙΕΔ. Δεν έχω υπόψη μου τα ακριβή στοιχεία. Σήμερα αριθμούμε περίπου 100 άτομα στο Σίτσεν. Και όπως είπα, εξελίσσονται οι εργασίες μας ακόμη για να κάνουμε μια ανακατανομή των πόρων στο μέλλον και για να δούμε πόσο οι δραστηριότητες της ανταπόκρισης στην κρίση που διεξάγουμε στο πλαίσιο του, της διεύθυνσης της σχετικής, να δούμε πώς αυτό θα επηρεάσει και το ρόλο μας και το προσωπικό μου. Αλλά είμαστε γύρω στους 100 Τώρα, αν τα κράτη-μέλη απευθύνονται σε εμά και μα θέτουν ερωτήματα, πράγματι γίνεται αυτό. Ενίοτε ανταλλάσσουμε απόψε με τα κράτη-μέλη. Και θα έλεγα βέβαια ότι αυτό φυσικά εξαρτάται και από το θέμα και από το πόσο συχνά ε, έρχεται ένα κράτος μέλος να μας ε, ζητήσει συμβουλή και από το μέγεθος του κράτους μέλους. Τα μεγαλύτερα κράτη-μέλη πιο σπάνια μας ζητούν τη συμβουλή μας, για να το θέσω έτσι. Τώρα, κατά πόσο μπορούμε να στείλουμε επιτόπου άτομα. Ναι, πράγματι το κάνουμε αυτό σε κάποιε αποστολέ, αλλά πάντοτε με απόλυτη διαφάνεια. Δεν κάνουμε τίποτε στα κρυφά. Πάντα λέμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Αυτή είναι πολύ σαφής πολιτική γραμμή. Το έχω καταστήσει σαφές και στους υπαλλήλους μου ότι έτσι πρέπει να προχωρούμε. Και αν κάποιος πηγαίνει σε αποστολή, θα είναι διερευνητική αυτή η αποστολή Απλά δηλαδή συλλέγουν πληροφορίες με πολύ ανοιχτό τρόπο, όπως οποιοδήποτε άλλος υπάλληλο Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε. Κύριε Πρόεδρε, διαρωτώ με αν υπήρξαν ερωτήσεις οποίε ε, παρέλειψα να απαντήσω και αν το έχει συμβεί αυτό ευχαρίστω να το κάνω στη συνέχεια. Ε, μία τελευταία ερώτηση και Συγγνώμη, αν δεν κατάλαβα καλά, οι τρίτες χώρες. Διότι οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευαίσθητες περιοχές που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή από τις υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν όλο ένα και περισσότερο τρίτες χώρες ας πούμε με τη Σουή, με την Ελβετία ή την Νορβηγία δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν προβλήματα συνεργασίας για τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών αλλά με άλλες χώρες, άλλες τρίτες χώρες μπορεί να έχουμε πρόβλημα. Τώρα για το πρωτόκολλο το ΣΥΤΧΕΝ είναι ανοιχτό, το ΣΥΤΣΕΝ είναι ανοιχτό σε όλες τις συνεργασίες ο κύριος Ερνχάουζερ θέλει πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Ένα, μια αποφασιστική σημασία σε ερώτηση είναι πού ξεκινάει η δική σας υπηρεσία ή τέλος πάντων από πότε είναι λειτουργική η δική σας η υπηρεσία. Ε, είπατε ότι για τον παρακοινοβουλευτικό έλεγχο, εντάξει, μπορεί να μην είσαστε εσείς απόλυτα ε, απαραίτητοι, να μην είναι δηλαδή η δική σας υπηρεσία λειτουργική αλλά επειδή συνεργάζεστε και με τις αντιπροσωπείες και τα λοιπά, ε, συνεργάζεστε και με το κέντρο το δορυφορικό και τώρα μας είπατε ότι το προσωπικό σας επίσης πηγαίνει για επιτόπου ε, εξυχνίαση των, ε, της κατάστασης στις διάφορες περιοχές. Εσείς τα όρια που τα βάζετε, από πότε και μετά είναι επιχειρησιακή η δική σας υπηρεσία και από πότε δεν είναι. Και επίσης, για το τεχνικό, ε, το τεχνικό σύστημα με το οποίο δουλεύετε. Οι πληροφορίες πώς ανταλλάσσονται με τα κράτη-μέλη, δηλαδή τι τεχνικό σύστημα έχετε και ποιο είναι το τεχνικό σύστημα το οποίο επεξεργάζεστε. Ε, νομίζω το ΣΟΥΙ είναι αυτό που ε, ήδη έχει εφαρμοστεί. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε δύο πράγματα και γι' αυτό. Ευχαριστώ. Αυτά είναι τα δύο τελευταία σημεία. Mm. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την συνεργασία και τη μεθοδολογία. Σε σχέσεις εκτός ε, ένωσης είμαστε τώρα προσεκτικοί με ποιον θα συνεργαστούμε ή όχι. Και βέβαια η εφετηρία να έχουμε συμφωνία ασφαλείας με αυτό το φορέα, αν είναι διεθνής οργανισμός ή κάποιο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο τρίτο κράτος. Αυτή είναι η αφετηρία μας. Σήμερα εστιάζουμε κυρίως στη συνεργασία εντός πλαισίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έλεγα. Είπα και για την ε, Ελβητία και την ε, Νορβηγία ότι είναι στο πλαίσιο της αντικρομοκρατικής ομάδας ε, που εκεί περιλαμβάνονται και όλα τα άλλα κράτη-μέλη, όλα μάλλον τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα συνεργαζόμαστε στον τομέα του ΣΥΤ e με αυτές τις δύο χώρες και έχουμε και συμφωνία ασφαλείας μαζί τους. Επίσης, ε, διερευνούμε το ενδεχόμενο ανταλλαγής πληροφοριών με στρατηγικού επίπεδου αναλυτικούς οργανισμούς φορείς ανάλυσης ε, σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά αυτό είναι ακόμα υπό ανάλυση. Πρέπει να θεσπιστούν σαφέστατοι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Γιατί επανέρχομαι στο θέμα της εμπιστοσύνης που έχουμε με τους παρόχου πληροφόρων και τις υπηρεσίες των κρατών μελών. Επιχειρησιακό και στρατηγικό. Πώς θα όριζα αυτές τις δύο έννοιες. Ε, νομίζω ότι είναι και ενδιαφέρον το ερώτημα, αλλά είναι και σχετικά σαφής η απάντηση. Εγώ περισσότερο από ήθελα ήμουν στον τομέα των επιχειρήσεων και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ε, διάκριση μεταξύ ΣΥΤΣΕΝ και επιχειρησιακού οργανισμού, επιχειρησιακού φορέα. Εμείς δεν κάνουμε καμία μυστική υπηρεσία όπως σας είπα. Ούτε χρησιμοποιούμε μέσα εξαναγκασμού, ούτε χρησιμοποιούμε ανθρώπους ε, πληροφοριοδότες, δεν προσλαμβάνουμε πράκτορες, ε, δεν ε, διοικούμε πράκτορες και νομίζω ότι απέχουμε πόρο αυτού. Και θέλουμε να είναι πολύ σαφής η διάκριση επιχειρησιακό τακτικό αφενός, επιχειρησιακό ε, στρατηγικό μάλλον αφετέρου. Και ούτε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Ούτε και το κάνουμε. Και είναι και πιο στρατηγικές οι αναλύσεις μας. Όχι για το κατά πόσον αύριο θα υπάρξει ε, ένα σχέδιο τρομοκρατικής επίθεσης, συνωμοσία κτλ. Ή την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα για τα τεχνικά συστήματα μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και ημών. Οι υπηρεσίε των κρατών μελών χρησιμοποιούν τα δικά του συστήματα, άρα έχουμε πολλά συστήματα. Φαντάζομαι ότι δεν θα χαίρονταν και πολλοί οι υπηρεσίε αν τα κατονόμαζα αυτά τα συστήματα. Και δεν με ενδιαφέρει καν, θα έλεγα. Εμένα με ενδιαφέρει το τελικό αποτέλεσμα, ότι υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών. Πάντως τα συστήματα τα παρέχουν οι υπηρεσίες οι ίδιες. Και έτσι έχουμε και την προστασία και τηρούνται και οι προδιαγραφές και οι απαιτήσει των υπηρεσιών των κρατών μελών. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για τις τοποθετήσεις Ελπίζω, όπως το επισήμανε και η κυρία Άγκης, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε γύρω από αυτό το θέμα. Δεν θα είναι πολύ ευτυχής οι συνάδελφοι της ΛΥΜΠΕ γιατί σε αυτό το τομέα υπάρχουν και θέματα άμυνας και ασφάλειας. Και όπως εσείς αναφέρατε δεν εργάζεστε ως μυστική υπηρεσία, δεν εργάζεστε παράνομα και δεν καταναγκάζετε. Θεωρούμε λοιπόν ότι η υποεπιτροπή μας θα συνεργαστεί στενά μαζί σας, τουλάχιστον θα σας συναντούμε. Συμμετείχαμε στην Ουγγάντα με ορισμένου συναδέλφου σε μία αποστολή όπου είχαμε πληροφόρηση ε, στην οποία και το ΣΕΤ ήταν αναμειγμένο. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Πέρα στη συνεδρίαση. Επόμενη συνεδρίαση την 5η 6 Οκτωβρίου.